Good morning, Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την ακρόασή μας για τον πλουραλισμό και την ελευθερία των ΜΜΕ στην Ένωση. Έχουμε μόνο δύο ρίτσες. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι θα έρθουν και άλλοι βουλευτέ, ελπίζω. Ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, όσου ήρθαν εγκαίρω. Δύο ώρες ε, είναι νομίζω ελάχιστος χρόνος για ένα θέμα τόσο μεγάλης σημασίας και το γενικότερο πλαίσιο έχει σημασία. Βλέπουμε δραματικές αλλαγές στον ε, τομέα αυτών και με χαρά καλωσορίζουμε τους ε, βουλευτές μας ε, και κυρίως την εισηγήτρια την Μπάρμπαρα Σπινέλη που θα μας μιλήσει σε λίγο ε, η Μπάρμπαρα έχει αναλάβει την έκθεση για τον πλουραλισμό και την ελευθερία των ΜΜΕ στην ε, ΛΥΜΠΕ. Η σημερινή μας ε, συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο, στον έξω κόσμο. Να πω δύο λόγια πριν δώσω τον λόγο στην Μπάρμπαρα. Οπότε αυτό το οποίο αποκαλούμε ελευθερία τύπου είναι μέρος των δημοκρατικών ιδεών και της εξέλιξης του ευρωπαϊκού ιδεώδους σε ολόκληρη την ιστορία. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν και σημασία και για τους βουλευτές μας. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η ελευθερία των ΜΜΕ είναι ένα κριτήριο για την ένταξη οποιασδήποτε υποψήφιας χώρας, σύμφωνα με την κριτήρια της Κοπενχάγης. Είναι λοιπόν πολύ βασικό για εμάς και την νομική μας βάση. Είναι μία από τις αρχές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξωτερική της πολιτική και ενώ τα κράτη-μέλη βεβαίως θα πρέπει να ηγούνται δια του παραδείγματος. Βεβαίως ε, τα πράγματα αλλάζουν ε, μέσα στον χρόνο και η ακρόαση σήμερα έχει σκοπό να καθορίσει το τι εννοούμε ελευθερία των ΜΜΕ. Θα ακούσουμε λοιπόν σήμερα τους ειδικού για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και για να γίνει αυτό πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τους ε, εισηγητές μας ε, και μια σειρά ειδικών. Επίσης έχετε μια μελέτη που προετοιμάσαμε, ένα τμήμα της ανάλυσης ε, που κάναμε, που έκανε το τμήμα πολιτικής, που έχετε όλοι. Έχουμε λοιπόν και την, για να βοηθήσει και την εισηγήτρια και την σημερινή συνεδρίαση. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα δώσω τώρα τον λόγο στην εισηγήτρια για να μπούμε στην ουσία τη σημερινής ακρόασης. Κυρία Σπινέλη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ και τους, εισηγή, τους ε, εμπειρογνώμονες που θα πάρουν το λόγο στη διάρκεια του της, της ακρόασης. Ως εισηγήτρια μιας νέας έκθεσης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης σας, ε, σας λέω εξ αρχής ε, ότι θα είναι πολύτιμη η συμβολή σας θέλουμε να καταλήξουμε σε μια εργασία στην οποία ε, ε, στην ε, μελλοντική μας έκθεση θα εισάγουμε και στοιχεία τα οποία θα αποκομίσουμε από σήμερα. Εγώ επί δεκαετίες δούλευσα ως δημοσιογράφος και πλέον η κατάσταση είναι ιδιαίτερος δύσκολη. Η, η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων είτε από οικονομικό κέντρα ενδιαφέροντος ε, είτε ε, από τις ε, πολιτικές ε, αρχές ε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μάλιστα έχει δυσκολέψει, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση από το 2013 που ήταν η τελευταία φορά που το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αφήσω όλο το δυνατό χρόνο για τους εμπειρογνώμονες αλλά θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι η κατάσταση είναι αρρωστημένη παντού. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία ε, στα οποία ε, οφείλεται η επιδείνωση και κατά την άποψή μου θα πρέπει ε, να τα μελετήσουμε σε βάθος. Πρώτα απ' όλα τα fake news. Σε όλο και περισσότερες δημοκρατικές χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο, ο όρος αυτός κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης. Μερικοί μιλάνε για τα αλήθεια για, και αυτού του είδους τα νέα διευκολύνονται περισσότερο από τη χρήση των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε το την γέννηση των fake news, να χτυπήσουμε την ρίζα τους και κυρίως ε, να ε, προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε από αυτά τα fake news ε, τον χώρο του διαδικτύου. Γιατί αυτά τα fake news δεν είναι ακριβώς ασθένεια του διαδικτύου, είναι μια ασθένεια η οποία ξεκίνησε από, την, από τις, το γραπτό τύπο και τις εφημερίδες ως κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου. Ε, εκεί, από εκεί ξεκίνησαν αυτές οι ψευδείς ε, ειδήσει ε, και ας πούμε κανείς μπορεί να σκεφτεί αυτές τις ψευδείς ειδήσει σχετικά με το πυρηνικό πλωστάσιο και το, και το προστάσιο γενικά του Ιράκ. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τις ειδήσει κυρίως κυρίως όταν προέρχονται από μεγάλα μέσα ε, και ε, βεβαίως είναι μια προσπάθεια να φημωθούν εν τέλει τα μέσα ενημέρωσης ξεκίνη, έχει μακρά ιστορία η δημοσιογραφία ε, και από αρχής ε, της, ε, της δημοσιογραφίας, γραπτής, ραδιοφωνικής κλπ. η προσπάθεια καταστολής της ελευθερίας είναι συγκεκριμένη και διαρκής. και από την άλλη πλευρά βεβαίως το να λέει ο καθένας ό,τι θέλει τελικά είναι αντιπαραγωγικό. Η υπερβολική δημοκρατία εν τέλει σκοτώνει τη δημοκρατία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τις ε, ε, ρίζες λοιπόν του ε, κακού. Αυτό ήταν το πρώτο μου σημείο. Δεύτερο ε, πρόβλημα είναι η επέκταση ε, παλαιών φαινομένων που όμως ε, όχι μόνο διαρκούν αλλά και αυξάνονται. Η παρέμβαση της πολιτικής, η βία κατά των δημοσιογράφων, ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων και των πληροφοριοδοτών τους αλλά και οι πολλοί διάχυτες τις ε, και διαδεδομένες πλέον ε, πρακτικές αυτολογοκρισίας. Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι πιέζονται έτσι ώστε να μην αποκαλύψουν όλη την αλήθεια ε, και αυτό είναι μια παθολογία η οποία ήδη εφήγει στην προηγούμενη έκθεση του Κοινοβουλίου αλλά δεν μελετήθηκε σε βάθος. Δεν μελετήθηκε δηλαδή ο μηχανισμός ο οποίος οδηγεί στην αυτολογοκρισία ή πολλαπλασιασμός των ε, μεθόδων ε, που χρησιμοποιούν οι κέντρα εξουσίας έτσι ώστε να προκαλέσουν φόβο, να εκφοβήσουν ε, και έτσι ώστε ο δημοσιογράφος πλέον όπως και οι πληροφοριοδότες να βρεθούν σε όλο και πιο δυσχερή θέση. Η πραγματική ρίζα των ψευδών ειδήσεων όπως και αυτή της αυτολογοκρισίας δεν αποκαλύπτεται και νομίζω ε, ότι είναι ε, αυτή η έκφραση ενός ε, ορθολογικού κομφορμισμού που επιβάλλεται από ομάδες οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ο William ε, ο οποίος δημιούργησε τον όρο τη δεκαετία του 50, ε, λέει ότι είναι μια φιλοσοφία δεδηλωμένη και διαρθρωμένη η οποία ε, θεωρεί ότι οι αξίες των ομάδων δεν είναι μόνο καλές αλλά είναι και σωστές ο όρος τώρα απλώς έχει εκσυγχρονιστεί. Τρίτο σημείο, αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο, είναι σημαντικό θέμα στις Δημοκρατίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίλημα της Κοπενχάγης οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες ε, πρέπει να σέβονται ε, τις ε, αρχές της ελευθερίας του τύπου, της ελευθερίας του λόγου και τα όσα αναφέρονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κυρίως δε τα άρθρα 10 και 11. Αλλά όταν εισέρχονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι όλα επιτρέπονται. Την τελευταία δεκαετία έχουμε δει, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία. Έχουμε δει συγκεκριμένες παρεμβάσεις ε, στο δημοσιογραφικό έργο. Θεωρώ ότι ε, ε, στην ε, χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφέρεται όμως αφώς και, η, και ο πλουραλισμός των μέσων. Τέλος το θέμα των πληροφοριοδοτών. υπάρχουν δύο άρθρα που αφορούν την νομική προστασία των πληροφοριοδοτών αλλά λείπει η αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες τιμωρητικές μακρές διαδικασίε οι άνθρωποι αυτοί. Επομένως είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη ένταση. Πέμπτο σημείο αφορά ε, τις επιπτώσεις της οικονομικής ε, κρίσης ε, η οποία αυτή η οικονομική κρίση έχει ε, στο εσωτερικό της ε, και μία κρίση των μήνυ ε, ε που αφορά πλέον και την ίδια την ύπαρξή τους. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι έχουν ήδη προβλέψει την ημερομηνία θανάτου του χάρτινου του έντυπου τύπου οι πληροφοριοδότες και οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι βρίσκονται όλο και σε πιο δύσκολη θέση γιατί ε, στην ουσία βρίσκονται στο έλεος ε, μιας ε, πολύ μικρής ομάδας παλαιών αρχών δημοσιογράφων ενώ πληθαίνουν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι δουλεύουν είτε με εξευθελιστικούς μισθούς είτε και δωρεάν. Θα πρέπει να οργανωθούν καλύτερα οι δημοσιογράφοι να προσαρτηθούν στην χάρτα των δικαιωμάτων και επομένως να έχουν σωστή αμοιβή. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στη σύμβαση και πιστεύω ότι άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρομαι στην έκθεση της Εσόφη Ίντβελτ του προηγουμένου Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύτιμο ακριβώς διότι ε, ενέχεται σε αυτήν ε, και η κοινωνία των πολιτών. Επομένως, ε, ε, αυτό περιμένουμε ε, και από σας να μιλήσετε και για αυτό το θέμα, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης πριν από την προσφυγή τύπου του άρθρου 7 και που επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς λόγω του προκεχωρημένου σταδίου στο οποίο καλείται να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ Μπάρμπαρα, λέει ο Πρόεδρος. Με τον τρόπο αυτό κατανοήσαμε και τη δομή της έκθεσής σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Έχουμε τέσσερις ε, καλεσμένους. Ε, να παρακαλέσω όλους τους ομιλητές ε, να μην υπερβούν τα δέκα λεπτά. Ξέρω ότι το αντικείμενο είναι τέτοιο που θα μπορούσατε να μιλάτε επί ώρες, αλλά παρακαλώ να μην ξεπεράσετε, να μην υπερβείτε τα δέκα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τον Πιέρ Λουίτζι Πάρκου ο οποίος ε, είναι επικεφαλής ε, του Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου. Ε, πρόκειται για ένα κέντρο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει μελέτες και έρευνες σχετικά με την ελευθερία και το πλουρισμό του τύπου. Έχει προσφάτως δε ο Πιέρ Λουίτζι δημοσιεύσει την τελευταία έρευνα για το 2016. Ευχαριστώ. Θα παρουσιάσω τα πορίσματα της ε, μελέτης μας για το 2016. Πρόκειται για ανεξάρτητη μελέτη όσον αφορά την πολυφωνία στον τύπο. Αξιολογούμε τον κίνδυνο για την πολυφωνία σε ένα κέντρο το οποίο, όπως είπαμε, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016 ήταν η πρώτη μας πλήρης ε, έκθεση. Ε, έχουμε 22 χώρες ε, έχουν επίση κάνει αίτηση, η Τουρκία και το Μαυροβούνιο. Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι η εξή. Αναλύουμε τέσσερις τομείς, τέσσερα αντικείμενα βάσει 200 περίπου ποσοτικών και ποιητικών παραμέτρων. Έχουμε 28 κρατόπους ομάδες εμπειρογνώμων, συν Ιταλία και Μάλτα που ε, εξετάζουμε κατευθείαν, κεντρικά δηλαδή από την ομάδα μας του CMPF. Χρησιμοποιούμε πρωτογενείς πηγές στοιχείων αλλά και δευτερογενείς. Έχουμε εμπειρογνωμονές παντού. Έχουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων που συγκρίνουν τα επιμέρους αποτελέσματα σε συνεργασία με τις κρατόπους ομάδες και καταλήγουμε στο τελικό πόρισμα. Για την συλλογή των δεδομένων έχουμε ένα διαδικτυακό εργαλείο, ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ακριβώ τον κίνδυνο λαμβάνοντα υπόψη και συγκεράζοντα πολιτικέ, οικονομικέ και άλλε παραμέτρου. Είναι το σύστημα των σηματοδοτών, τα τρία χρώματα όπω ε, γνωρίζετε. Δηλαδή έχουμε χαμηλό, μέσο και υψηλό κίνδυνο, κάπω έτσι μετράμε χρόνο διδάσκοντα των κίνδυνο, Να σα πω για τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Το 2016 λοιπόν έλεγα ο πρώτο τομέα που είναι και πιο σημαντικό είναι η βασική προστασία των θεμελιωτών, δηλαδή δικαιωμάτων ελευθερίας κλπ. Εδώ είναι σαφές ότι η Ευρώπη τα πηγαίνει σχετικά καλά, έχουμε νομοθεσία, έχουμε θεσμούς, παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Ο βασικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος για τα παραδοσιακά μέσα εν ώψη της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσος κίνδυνος και δεν έχουμε ικανοποιητική κατάσταση στα δικαιώματα πρόσβαση στο επάγγελμα κλπ. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη. Η μόνη χώρα με κόκκινο είναι η Τουρκία. Και αυτό μάλιστα πριν το πραξικόπημα, οπότε έχετε μια ιδέα. Θα επανεξετάσουμε φυσικά την Τουρκία και φέτο, αλλά ε, θα δούμε τι έγινε μετά το πραξικόπημα, όπου τα πράγματα είναι σίγουρα χειρότερα σε σχέση με πριν. Έχουμε κίτρινο σε διάφορε άλλε χώρε. Ε, μετά, πολυφωνία της αγοράς. Εδώ μελετούμε την συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων και τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα, εν προκειμένου, ε, είναι εδώ φαντάζεστε λιγότερο καλά. Το χειρότερο αποτέλεσμα, χειροτερή βαθμολογία, αφορά τη συγκέντρωση των μέσων, τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας. Θα πάμε καλύτερα ε, στον έλεγχο του περιεχομένου και εδώ όσον αφορά την αυτονομία των ε, συντακτών κλπ. Έχουμε μέση προστασία. Προστασία εργαζομένων και συντακτών από την ιδιοκτησία. Εδώ η Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο είναι στο κόκκινο. Το Λουξεμβούργο βεβαίω είναι μικρή χώρα και πρέπει να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει το κόκκινο για το Λουξεμβούργο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά κίτρινα, αυτό είναι το ανησυχητικό, όπου η πολυφωνία λοιπόν της αγοράς του τύπου αξιολογείται ως μέσο κινδύνου. Τρίτος τομέας, πολιτική ανεξαρτησία. Εδώ αξιολογούμε την πολιτικοποίηση του συστήματος, την οργάνωση των μέσων σε μια χώρα, την αναφορά των νέων, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια μέσα κλπ. Εδώ έχουμε ψηλού κινδύνου, Οι δύο δείκτε που προκαλούν περισσότερη ανησυχία είναι ο πολιτικό έλεγχο των μέσων. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε καθημερινά. Σε πολλέ περιοχέ είμαστε κοντά στο κόκκινο, υπάρχει υπερβολικά πολύ πολιτικό έλεγχο κάτι το οποίο θίγει την αυτονομία των συντακτών. Και αυτό φαίνεται και στον επόμενο δείκτη. Δεν προστατεύεται παρκώ η ανεξαρτησία των συντακτών από πολιτικέ παρεμβάσει. Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα. Και αν πάμε στο χάρτη, και πάλι ως αναμένεται η Τουρκία είναι στο κόκκινο, αλλά βλέπουμε και το Μαυροβούνιο, είναι προβληματικό και βλέπουμε επίσης σε κόκκινο τη Σλοβενία αλλά και την Ουγγαρία. Μερικέ κίτρινες χώρες είναι πολύ κοντά στο κόκκινο πρέπει να σας πω, αλλά ήδη είναι ανησυχητικό το ότι έχουμε πολλά κίτρινα. Ε, το καλό είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στο πράσινο. Τεταρτο δείκτη, κοινωνική συμπερίληψη. Δηλαδή, τι γίνεται με τα ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας, τι γίνεται με τις μειονότητες, τοπικές κοινωνίες, ε, γυναίκες, ε, άνθρωποι με αναπηρίες κλπ. Πώς τους μεταχειρίζεται ο τύπος. Και εδώ το αποτέλεσμα δείχνει ότι υπάρχουν μη ικανοποιητικές καταστάσεις ούτως υπήν, Τα χειρότερα αποτελέσματα είναι, αφορούν την πρόσβαση στα μέσα για τις μειονότητες. Εντυνόμενο πρόβλημα πρέπει να πω και το ίδιο ισχύει για μειονότητες που είναι αναγνωρισμένες αλλά και ακόμα χειρότερα τα πράγματα είναι για τις μη αναγνωρισμένες. Θα συνεχίσουμε να προσέχουμε αυτόν τον δείκτη. Επίσης η πρόσβαση των γυναικών στα μέσα μας εξέπληξε αυτός ο δείκτης. Ήταν η πρώτη φορά που μετρήσαμε αυτόν τον δείκτη σοβαρά και εξεπλάγημενο όπω είπα έχουμε εδώ μέσο κίνδυνο αλλά προς υψηλό. Αν πάμε ξανά στον γνωστό χάρτη θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Η Ελλάδα είναι επίσης εδώ στο κόκκινο και η Λετωνία. Και πάλι όμως πολλά κίτρινα, αυτό είναι το ανησυχητικό, πολλές χώρες οι οποίες ε, δεν ε, παρουσιάζουν ικανοποιητική κατάσταση. Τα πράσινα δεν έχει τόσο το, το, πράσι, το, το πράσινο, ξέρετε, ε, είναι μάλλον μια μέση κατάσταση. Δηλαδή, σε κάποιο δίκτυο μπορεί να τα πηγαίνει πολύ καλά μια χώρα, αλλά άσχημα σε κάποιον άλλον. Αν δούμε δηλαδή σε μεγαλύτερο βάθο, θα δείτε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα χάρη στη μελέτη που βρίσκονται πραγματικά κίνδυνοι. Ε, Προφανώ το πράσινο, το κόκκινο και το κίτρινο δεν σα δίνουν ε, λεπτομερή εικόνα των κινδύνων. Εν κατακλείδη, ο μηχανισμός που παρακολουθεί της είναι ένα καλό εργαλείο το οποίο έχει επαληθευθεί, έχει δοκιμαστεί. Κάναμε δοκιμές πριν από το 2016 σε όλες τις χώρες. Κάναμε δύο δοκιμές επί δύο χρόνια. Ξεκίνησε με 9 χώρες, μετά με 18. Λοιπόν, το εργαλείο δουλεύει. Έχει αποδείξει την αξιοπιστία του και μας παρέχει πολλές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τα μέσα είναι προσβάσιμο στο κοινό, μπορείτε να το δείτε στον ιστοτοπό μας, ούτως ή άλλως, όπως είπα, σύγχρονα το δείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν από δημοσιογράφου, εμπειρογνώμονες, ερευνητές, πολιτικούς, ε, φοιτητέ, δημοσιογραφίες κλπ. για όποιον θέλει να μελετήσει το χώρο σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Από εκεί πέρα, πρόκειται για εργαλείο αποτελεσματικό παρακολουθήσει τη κατάσταση. Όπω είπα, είναι αξιόπιστο. Μα βοηθάει να κατανοήσουμε του πραγματικού κινδύνου και να αποκτήσουμε περισσότερε γνώσει σχετικά με το πού η κατάσταση είναι ενδεχομένω ανησυχητική και πού ενδεχομένω και πάλι απαιτείται πολιτική απάντηση. Θα συνεχίσουμε και το 18 βεβαίω. Και για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία από έτος σε έτος. Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του 2018. Δεν έχουμε εξασφαλίσει η χρηματοδότηση για το μέλλον. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Φέρει ένα χρήσιμο εργαλείο, σαν εργαλείο επίση έγκαιρη προειδοποίηση και σαν ένα σημάδι ανάγκη νομοθετική αλλαγή. Το θέμα είναι όπου υπάρχει έστω και υποψία κινδύνου, υπονοή κινδύνου, να μπορεί κανείς να μελετήσει καλύτερα και να επεμβαίνει εάν βεβαίως υπάρχει τέτοια ανάγκη. Οπότε αυτά προς το παρόν η κατάσταση όπως προείπα δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Ε, ελοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τους κινδύνους αυτούς και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το συντομότερο δυνατόν, ειδικά όταν αναφέρονται συγκεκριμένα προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η ανάλυση και η διαφάνεια θα ανεβούν και στο site μετά την συνεδρίαση. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, νομίζω έχετε την δυνατότητα, γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, τώρα περνάμε στον κύριο Τάις Μπέρμαν που είναι ο κύριος σύμβουλος αυτή τη στιγμή στο γραφείο του εκπροσώπου για την ελευθερία των ΜΜΕ στον ΑΣΕ και η δουλειά του ΑΣΕ έχει μεγάλη σημασία για τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πούμε εδώ για λόγους διαφάνειας πως ο Τάις ε, υπήρξε βεβαίω και επί σειρά ετών Ευρωβουλευτής. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ Κλοντ μεγάλη μου χαρά επιστρέφω εδώ και βλέπω παλιούς συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν δουλειά μετά την δημοσιογραφία αλλά και μετά την πολιτική. Ε, υπάρχει η ζωή. Λοιπόν, βρίσκομαι στην Βιέννη, στον ΟΑΣΕ, όπου έχουμε εντός του ΟΑΣΕ ένα ανεξάρτητο σώμα. Πρόκειται για το μόνο παγκοσμίω ανεξάρτητο φορέα παρακολούθησης των ΜΜΕ που είναι διακυβερνητικός. Αυτό γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο. Ο ΑΣΕ βεβαίως ε, αρχικά ε, ήταν ένας οργανισμός για διάλογο ε, στρατιωτικών ζητημάτων μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Αλλά μετά σκέφτηκαν ότι η ασφάλεια περιέχει πολύ περισσότερα ζητήματα από τα στρατιωτικά και βεβαίω ε, σχετίζεται και με άλλες διαστάσεις όπως η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών. Και αυτό σημαίνει πως όταν δεν υπάρχει πλουραλισμός ε, θα υποφέρει η κοινωνία ολόκληρη. Και έτσι ο ΑΣΕ πέρασε από έναν οργανισμό διαλόγου του ψυχρού πολέμου για τις όροφες στρατιωτικών συστημάτων στο να προστατεύει τις ελευθερίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε εκπρόσωπο για την ελευθερία των ΜΜΕ. Το γραφείο υπάρχει, υπάρχουν 15 άτομα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε δημόσιες δηλώσεις γιατί δεν υπάρχει εκπρόσωπος. Είναι ενδεικτικό αυτό για την παράλυση που υπάρχει μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, ότι δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας του ΑΣΕ, δεν υπάρχει Διευθυντής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκλογών δεν υπάρχει υπατός εκπρόσωπος για τις μειονότητες και κανείς δεν ξέρει πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βρίσκεται σε κόμμα ο ΑΣΕ θα έλεγα. Θα ήθελα να τονίσω τρία πράγματα τώρα. Τρεις προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι η ασφάλεια των δημοσιογράφων η οποία βλέπουμε ότι απειλείται, υπάρχει σαφής αύξηση σε απειλές, παρενόχληση και βία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα 57 κράτη-μέλη του ΟΣΕ. Ειδικά οι γυναίκες δημοσιογράφοι κινδυνεύουν. Μετά έχουμε την ψηφιακή μετάβαση που θα ήθελα να τονίσω. Πώς θα προστατευτεί δηλαδή η ελευθερία των ΜΜΕ, ειδικά ο πλουραλισμό στην γρήγορο αυτόν ψηφιακό μετασχηματισμό που σημαίνει τεράστιε αλλαγέ, οικονομικέ και τεχνολογικέ δυνατότητε επίση. Προσπαθούμε δηλαδή να διατηρήσουμε τον πλουραλισμό και την ποιοτική δημοσιογραφία, ειδικά στις περιοχές της υπαίθρου. Το τρίτο. Οι αρχές, οι κυβερνήσεις δεν σέβονται πάντα τις υποχρεώσεις τους. Αναζητούν τρομοκράτες ε, και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον εξτρεμισμό και καμιά φορά ενέχουν τα μήμια το θεμελιώδες δικαίωμα για την ελευθερία έκφρασης φαίνεται ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή πολύ ψηλή προτεραιότητα και σε κάποια κάποια μέλη της Ένωσης. Το πρώτο θέμα λοιπόν, η ασφάλεια των δημοσιογράφων. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την αύξηση στις άπειλες ε, ε, παρενοχλήσεις, εκφοβισμούς ε, δημοσιογράφων. Εκφύσεως εξορισμού είναι πολύ ορατοί άνθρωποι, υπάρχουν εκεί όπου υπάρχει ένταση στην κοινωνία, αναλύουν διλήμματα και γνώμες. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολη στόχη. Στην Ολλανδία, στη χώρα μου, 62% των δημοσιογράφων έλαβαν, δέχτηκαν απειλές πέρσι. Και από τις αρχές. Του λένε π.χ. θα σας κάνουμε μήνυση άμα το δημοσιεύσετε. Ή απειλές ε, θανάτου, βιασμού κτλ. Οι γυναίκε δημοσιογράφοι υφίστανται τη χειρότερη πίεση και είναι με προτεραιότητά μας. Ε, εκδώσαμε και μία έκθεση δηλαδή. Η χαρακτηριστική αντρική επιθετικότητα ε, των ανδρών απέναντι στις γυναίκες προστίθεται βεβαίως ε, στον μίσο κατά των δημοσιογράφων και πολλοί πολιτικοί λένε ότι τα ΜΜΕ είναι εχθρό του λαού. Οι απειλέ αυτές έχουν σοβαρέ συνέπειε για την ποιότητα του δημοκρατικού διαλόγου γιατί οδηγούν σε αυτολογοκρισία. Πριν ε, δημοσιευθεί π.χ. ένα θέμα για την άκρα δεξιά ή άλλες δήματα, οι αρχείς κατά κανόνα αναρωτιούνται αν αξίζει τον κόπο και ξέρουν και είναι πολύ σημαντικό αυτό Ε πρέπει να τονίσουμε αυτό ξέρουν ότι οι ιδιοκτικές αρχές δεν ασχολούνται τώρα με αυτά τα θέματα οι ιδιοκτικές αρχές γενικά δεν δρούν ε, για ε, απειλές και εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η αυτολογοκρισία δεν είναι προς το συμφέρον των δημοκρατιών δεν θα βρεθούν με το να κρύβουμε τα γεγονότα. Η δημιουργικότητα μιας κοινωνίας εξαρτάται από μια ανοιχτή ατμόσφαιρα. Οπότε χρειάζεται μια δέσμευση της Ένωσης πως οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων δεν θα γίνουν ανεκτές. Και θα πρέπει να υπάρχει κάποια παρακολούθηση από τις διοκτικές αρχές. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπαμε, εκτίθενται ε, όπως και η αστυνομική. Δεύτερον, η ψηφιακή μετάβαση. Το Facebook και το Google είναι πλέον οι παγκόσμιοι αρχισυντάκτες και έχουν σχεδόν 80-85% του ε, διαφημιστικού εσόδου στο διαδίκτυο. Έτσι υπάρχει μια συγκέντρωση των ΜΜΕ με ένα τεράστιο αντίκτυπο στον πλουραλισμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε ένα τέταρτο ή και σε ένα τρίτο των ε, δήμων ε, των, ε, της περιφέρειας δεν υπάρχουν ανεξάρτητα έντυπα, χάρτινα έντυπα. Δεν υπάρχει επίση κάποιο ανεξάρτητο έλεγχο των τοπικών αρχών. Όχι μόνο στον Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, την Ολλανδία. Δηλαδή συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια χωρίς παρουσία δημοσιογράφων, εντάξει τα blog και τα λοιπά καλά είναι, αλλά δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν αυτό. Επίσης ε, έχει εξασθενήσει η οικονομική θέση των χάρτινων εντύπων, των εντύπων. Είναι παράδοξο του διαδικτύου το ότι κάθε πολίτης έχει γίνει πιθανή πηγή πληροφόρησης, κάτι το οποίο βεβαίως έχει οθήσει πολύ τον δημοκρατικό διάλογο, αλλά ο πλουραλισμό και η ποιοτική δημοσιογραφία κινδυνεύουν. Η ανεξαρτησία των ΜΜΕ κινδυνεύει. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να παίξει να δημιουργήσει κάποια σαφήνεια όσον αφορά τις επιλογές δημόσιας χρηματοδότησης των ΜΜΕ, αλλά και ακόμα περισσότερες επιλογές για να διευκολυνθεί ο διάλογος για κάποια βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα το τμήμα πολιτικής ε, του Κοινοβουλίου έβγαλε μια εξαιρετική έκθεση που υπάρχει στην ε, είσοδο της αίθουσας που τονίζει τις δυσκολίες των ΜΜΕ και ειδικά τις απαράδεκτες πολιτικές πιέσεις σε κάποιες χώρες. Το τρίτο. Δεσμεύσεις, υποχρεώσει και πραγματικότητα. Κάποιες κυβερνήσεις ε, έχουν τον πειρασμό του να επανέλθουν στην παλιά και γνωστή οδό της λογοκρισίας για να καταπολεμήσουν την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Όχι, πρέπει να αποκαλύπτουμε τα ψέματα, τις φήμες, τις ψευδεί ειδήσει, οπότε χρειάζεται περισσότερο ποιοτική δημοσιογραφία. Και πολλές ποιοτικέ εφημερίδες ε, του θεωρούν προτεραιότητά του αυτό. Το ίδιο κάνει βεβαίως και η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσει, αλλά αυτό αφορά μόνο τι πληροφορίε που εκπορεύονται από τη Μόσχα. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, π.χ. ψευδέι ειδήσει που διασπείρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα χώρε μα. Ε, τον Μάρτιο, ο εκπρόσωπό μα η η μα μας κυρία Μιάτοβιτς ε, εξέδωσε μια δήλωση για τις ψευδείς ειδήσει και την παραπληροφόρηση μαζί με τους εταίρους της από τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και την Αφρικανική Ένωση. Και η σύστασή τους είναι όχι λογοκρισία, έρευνα, αποκάλυψη και βεβαίως να αυξηθεί περισσότερο η ενημέρωση γύρω από τα μήμια. Οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις επίσης έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν καθώς δεν εξαρτώνται από εμπορικά συμφόρτα και είναι ενισχυτικό ότι μια χώρα όπως η Πολωνία έχει θέσει τα δημόσια μημία υπό αυστηρό κυβερνητικό έλεγχο η εκπρόσωπος μας ε, άσκησε κριτική σε αυτόν τον νόμο και παρακολουθούμε ότι απολύθηκαν πάνω από 200 δημοσιογράφοι είτε μετατέθηκαν είτε αναγκάστηκαν να παρέτηθούν. Δυστυχώς κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες δεν πρέπει να τους εμποδίζουν να κυνηγούν τρομοκράτες. Αυτό ξεκίνησε βεβαίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου και δεν έχει τελειώσει. Η υπηρεσία μας έχει προειδοποιήσει γι' αυτό. Δεν έχει νόημα να σκοτώνουμε τι ελευθερίε για να τι σώσουμε. Οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τι πηγέ του. Η μαζική παρακολούθηση θα πρέπει τουλάχιστον να εξαιρεί τι επικοινωνίε μεταξύ δημοσιογράφων και των πηγών του. Η Ολλανδία είναι μια χώρα όπου το βασικό αυτό δικαίωμα των δημοσιογράφων δεν προστατεύεται ε, στον νέο νόμο περί υπηρεσιών ασφαλείας. Ε, θέσαμε το ζήτημα, δυστυχώς χωρίς επιτυχία. Οι νόμοι περί ρητορικής μίσους επίσης περιορίζουν ελευθερία του λόγου, όπως στη Γερμανία, και επίσης υπάρχουν δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα που οδηγούν σε προληπτική λογοκρισία από το Facebook, αλλά τα όρια πρέπει να καθορίζονται εκ των υστέρων και όχι πριν εκφραστεί ένας πολίτης και μόνο από δικαστές. Τέλος, η δυσφήμιση εξακολουθεί να υπάρχει στον ποινικό κώδικα των περισσότερων κρατών μελών. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να πάνε στη φυλακή, θεωρητικά. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό έχει ζητήσει η υπηρεσία μα επί σειρά ετών, αλλά η αλλαγή είναι πάρα πολύ αργή. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Μάλτα. Άλλαξε τον νόμο περί δυσφήμιση και ΜΜΕ κατόπιν σύμβουλων μα και πλέον η δυσφήμιση δεν είναι ποινικό αδίκημα. Α, έχω ξεπεράσει το χρόνο. Να σα δείξω τον χάρτη στο κόκκινο βλέπετε τις χώρες όπου εξακολουθεί να υπάρχει δυσφήμιση στον ποινικό κώδικα. Οι περισσότερες χώρες δεν εφαρμόζουν ποινές, αλλά θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να αποποινικοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει μοντέλο για την ελευθερία των ΜΜΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω ότι ε, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να υποστηρίξουμε τους ε, δημοσιογράφους, την φυσική τους και πνευματική τους παρουσία. Ναι, βεβαίως είσαστε παλαιός βουλευτής, ήταν λογικό και αυτονόητο ότι θα ξεπερνούσατε το χρόνο ομιλία σας. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα ε, να ε, δώσουμε τον λόγο στον ε, εκπρόσωπο των δημοσιογράφων. Παρακαλώ. Thank you very much. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Λίμπε που ε, διοργάνωσε αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ευχαριστώ βεβαίως και την Μπάρμπαρα Σπινέλη ε, η οποία έχει τόσο αυτό το βάρος να παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Εμείς εκπροσωπούμε 40 οργανώσεις ε, στα πλαίσια των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω ε, για, τον, για την έκθεση για τον ε, πλουραλισμό των ε, μέσων ε, που εκπονείται από το Κέντρο για την Πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης. Είναι η έκθεση αυτή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό εργαλείο που θα πρέπει να μοιράζεται παντού. Ήμουν πρόσφατα στην Ιρλανδία όπου η συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης έχει λάβει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις ήρθαμε σε επαφή ε, με ε, πολλούς δημοσιογράφους αλλά και με πολιτικούς και προς ώρας έχει σταματήσει η συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης. Ε, οπωσδήποτε ε, συμμεριζόμαστε το συμπέρασμα ότι η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης μπορεί να αποτελέσει πρόσκομα ε, στην πληροφορία και την πολυφωνία και ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ξεκίνησα πριν από 25 χρόνια και ε, ε, άσκησα πίεση ως λόμπιστε για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Ε, βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά έχει προωθήσει τα θέματα αυτά, αλλά τα κράτη-μέλη εν τέλει είναι αυτά τα οποία τότε δεν είχαν πάρει πολύ συγκεκριμένη θέση και ισχυρή θέση απέναντι στο τον τότε και αντίστοιχες ε, ε, περιπτώσεις. Η πράσινη βίβλος ε, για το θέμα αυτό δεν προωθήθηκε πολλέ, ποτέ και γι' αυτό προχώρησε η συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης και διονγκώθηκε το πρόβλημα. Είναι κατανοητό βεβαίως ότι το θέμα αυτό τώρα βρίσκεται στην κορυφή του πολιτικού θεματολογίου μαζί με τις ψευδείς ειδήσει. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά εάν δεν αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε ε, τα κύρια αίτια τα οποία οδηγούν στην αποτυχία εν τέλει ε, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης δεν θα καταφέρουμε και πολλά. Το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης είναι πράγματι περίπλοκο, αλλά η άνευ προηγουμένου συγκέντρωση ε, μέσων ενημέρωσης και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Εσείς μάλιστα κύριε Μπέργμαν αναφερθήκατε και στο καθαρά τοπικό επίπεδο. Εάν λέω δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και αν δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το διοκτησιακό καθεστώς, τότε δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση σε αυτό το ε, σημαντικό πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μια λύση ε, ε, και αυτή είναι η πολυφωνία. Βεβαίως είναι πιο εύκολο να το πει κανείς παρά να το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμούμε ιδιαίτερο τα όσα κάνετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Είδαμε μάλιστα χθε ότι και η Εστονική Προεδρία αύριο οργανώνει σεμινάριο για την πολυφωνία των μέσων και το κράτος δικαίου την ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ε, και είδα ότι και η Γενική Συνέλευση επίσης θα ασχοληθεί με αυτό το EFJ σε ένα ε, πρόσφατο ψήφισμα του Μαΐου στο, στην, ε, στο Βουκουρέστι αναφέρθηκε ε, στην απόφαση της Κομισιόν της 7ης Απριλίου του 2017 ε, ε, σχετικά με την ε, εξαγορά του Sky από, το, από την 21st Century Fox, δηλαδή του Mertok. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά και του περιεχομένου αλλά και των τηλεοπτικών σταθμών. Κατά την άποψή μας η Κομισιόν με την απόφαση αυτή δεν έλαβε υπόψη της τη δεσπόζουσα θέση του Murdoch Επίσης επίσης δεν έλαβε υπόψη και την επιρροή που μπορεί να έχει η Fox σε διάφορες ε, αγορές είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε αλλού. Και επίσης το γεγονός ότι ο Μέρντοκ Πολάκης έχει ξεπεράσει τα όρια ε, της ε, επιρροής του και ε, επίσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη ε, τα δικαιώματα ε, της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώθηκαν τα μονοπόλια του τύπου και επομένως μειώθηκε η πολυφωνία και η πολυμορφία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να σας, ε, να σας διαβάσω ε, κάποια στοιχεία από το περσινό ψήφισμα ε, του, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λέει, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής, μάλλον όχι, τα μέλη της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τροποποιήσουν το, το, τους τους έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια ε, πολυφωνία, να γίνει σεβαστή η πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω της, του περιορισμού ιδιοκτησιακού καθεστώτος που θα επιτρέπει δεσπόζουσα θέση. Αυτό λέει ότι, ε, ε, από μόνο του ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε καινούριε νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν ήδη οι κανονιστικές ρυθμίσεις, απλώς θα πρέπει να, γίνουν, να εφαρμοστούν και θα πρέπει να υλοποιηθούν Υπάρχουν ε, ήδη υφιστάμενα κείμενα, πράγμα που είπατε και εσείς κύριε Μπέρμαν προηγουμένως. Θα ήθελα τώρα να κάνω ε, κάποια σχόλια όσον αφορά το MPM, το οποίο ε, αναφέρεται προηγουμένως. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως όσον αφορά την προστασία των ε, ε, δημοσιογράφων. Είπατε κι εσείς ε, ότι τα, η προστασία των προτύπων του δημοσιογραφικού επαγγέλματος αλλά και η ίδια η ασφάλεια του δημοσιογραφικού επαγγέλματος είναι ένα ζητούμενο. Η Κροατία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Λετωνία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η Ουγγαρία και βεβαίως και η Τουρκία, αυτό δεν μας εκπλήσει. Οι χώρες οι οποίες μελετήθηκαν μας έδωσαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η στις περισσότερες από αυτές τις χώρες αναφέρονται προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Η ανάλυση των ε, δικτών ε, αναφέρει ότι, και συγγνώμη που επαναλαμβάνω, ότι ε, οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, φυσικές και ψηφιακές απειλές, λογοκρισία και υποχρέωση σε αυτολογοκρισία κλπ. Και τα στοιχεία αυτά ε, επίσης επιβεβαιώνονται από την πρόσφατα δημιουργημένη πλατφόρμα ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επομένως, ε, οι κυβερνήσεις ε, δεν έχουν καλύψει, δεν έχουν καταφέρει δηλαδή να καλύψουν ε, τις βασικές ανάγκες οι οποίες απαιτούν την σωστή συμμετοχή των δημοσιογράφων στη δημόσια συζήτηση. Και η επανειλημμένα έχει αναφερθεί το θέμα αυτό. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης πλέον έχουν γίνει κενό γράμμα, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ενταχθεί στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει και οι δημοσιογράφοι και όλοι όσοι εμπλέκονται στο δημοσιογραφικό επάγγελμα θα πρέπει να δουλεύουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει. Ευελπιστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει έτσι ώστε ε, να ε, σπρώξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να οθήσει, να πιέσει τις χώρες μέλη να προστατεύουν την δημοσιογραφία και τους ε, δημοσιογράφους. Ε, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόσφατο ψήφισμα το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ε, ομόφωνα πλην της Ρωσίας, έγινε δεκτό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, στην ίδια σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, προτείνεται η αναθεώρηση των εθνικών ε, νομοθεσιών όσον αφορά την ελευθερία του δημοσιογράφου και της, του δημοσιογραφικού επαγγέλματος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ανεξαρτησία. Η έκθεση, η εθνική, μια εθνική γενική έκθεση ε, αξιολόγησης ε, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του τύπου ε, θα έπρεπε να έχει συνεχθεί από όλες τις χώρες αλλά δεν έγινε ποτέ. Ένα άλλο σημείο το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό και αφορά την, ε, τους δημοσιογράφους και την εργασία τους ε, είναι οι συνθήκες ε, εργασίας. Το 2015 οι συνθήκες εργασίας συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση. Είναι ιδιαίτερε προβληματικές στη Λετωνία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και στην Τσεχική Δημοκρατία. Νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι πόσο πρόσκαιρη είναι η κατάσταση της, ε, ε, των ε, δημοσιογράφων και μάλιστα στο ενημερωτικό δελτίο του, των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχει, έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα πολλές περιπτώσεις burn-out, εξάντλησης λόγω υπερβολικής δουλειάς όπου στους δημοσιογράφους ε, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ε, διαδεδομένοι. Ε, οι δημοσιογράφοι, πολλοί δημοσιογράφοι δεν έχουν πλέον διάθεση να παραμείνουν στο δημοσιογραφικό επάγγελμα γιατί, αυτό, γιατί οι συνθήκες έχουν τόσο επιδεινωθεί. Και επίσης ε, υπάρχουν και αυτές οι περίφημες κατευθυντήριες γραμμές ε, ε, συστάσεις του Συμβουλίου που αναφέρουν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν σημασία εις τους εργατικούς νόμους και στην εργατική νομοθεσία έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η επισφαλής εργασία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους δημοσιογράφους. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η, ε, πολυφωνία ε, έτσι όπως ε, πρέπει να εμφανίζεται στον, στον τύπο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πλέον μία τάση για υπερβολικά μονοδιάστατη παρουσίαση το, των δημοσιογραφικών πληροφοριών και το σημείο αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη και την προσφυγική κρίση. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αναφέρω είναι ότι η ανάγνωση του τύπου είναι ε, πλέον ε, ε, ιδιαίτερα προβληματικό γεγονός. Είναι ένα στοιχείο το οποίο όμως πρέπει να βρίσκεται ψηλά στο θεματολόγιο. Πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνική ανεξάρτητη δημοσιογραφία θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε νέες ιδέες, ενδεχομένως να χρηματοδοτηθούν ε, πλατφόρμες όπου οι δημοσιογράφοι μπορούν ανεξάρτητα να γράφουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Νομίζω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Και τώρα η τελευταία εμπειρογνώμων, Μαρία Κλάρκ, επίκουρη καθηγητρία στην, ε, στην ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας ασκεί δημοσιογραφία υποπίεση. Συγχωρείτε, το θέμα της είναι δημοσιογράφη υποπίεση, τις παρεμβάσεις, φόβος και αυτολογοκρισία στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την, την πρόσκλησή μας. Θα ακούσουμε και μετά ερωτήσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στον πυρήνα της δημοκρατίας βρίσκεται το δικαίωμα της πληροφόρησης. Να δίνεις και να λαμβάνεις πληροφορία. Αυτό είναι προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε κοινωνίας, για την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας και κάθε ανθρώπου. Οι δημοσιογράφοι δραματίζουν προκειμένου πολύ σημαντικό ρόλο, κινούν τον δημόσιο διάλογο, ασκούν εποπτεία, ενημερώνουν για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, φροντίζουν για τη λογοδοσία των πολιτικών και για την επικοινωνία πολιτών με την εξουσία. Στα τελευταία χρόνια παρατηρούμε τακτικές με αντικείμενο, με σκοπό να σιωπήσουν οι δημοσιογράφοι. Έχουμε την σχετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου τονίζεται ότι πολλά κρατημέλη δεν εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον για τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι φυλακίζονται και μάλιστα σε αριθμούς χωρίς προηγούμενο. Αυτή η κατάσταση σοβεί εδώ και μία δεκαετία. Και ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο ε, καταρτήσαμε την μελέτη που θα σας παρουσιάσω. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε αξιόπιστα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα. Τρία βασικά ερωτήματα ερευνήσαμε. παρεμβάσεις, φόβος και σχέση μεταξύ αυτής της παρέμβασης του φόβου και της αυτολογοκρισίας. Ήταν μια έκθεση πρωτοβουλία ε, ο Τοσπίν με δείγμα περίπου χίλιους δημοσιογράφους από χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, άντρες και γυναίκες, Οι περισσότεροι είχαν μέση εμπειρία 16 έτη, 32% δούλευαν για εφημερίδες και κυρίως καλύπταν ε, θέματα κυβερνητικά. Μου ζητούσαν, ζητήσαμε από τους δημοσιογράφους μα μας από πού είναι. Καλύψαμε τρία χρόνια, όπως είπα, διάρκεια. Βλέπετε, μεγάλος αριθμός των απαντώντων είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τις άλλες χώρες. 24% από Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, 23% από Ανατολική Ευρώπη, 13% από Τουρκία και 6% από χώρες του Νοτιού Καυκάσου. Ιδού τα τεκμήρια που αποδεικνύουν αυτά τα οποία σας έλεγα. Βλέπουμε ότι Ανεπιθύμενες παρεμβάσεις είναι πολύ ψηλά. Ζητήσαμε από τους δημοσιογράφους να μας πούν τις εμπειρίες τους τα τελευταία ε, τρία χρόνια. Βλέπουμε ότι η ψυχολογική βία είναι πολύ ψηλά, 69%. Δύο τρίτα δηλαδή των δημοσιογράφων μας ενέφεραν ότι πέθαν ψυχολογική βία. Αυτό σημαίνει εκφοβισμό, περιφρονητική συμπεριφορά, παρενόχληση ε, και κυρίως από την εξουσία, όχι μόνο από τη διεύθυνση. Επίσης, ο εκφοβισμός, περίπου 50% μέσω διαδικτύου. Επίσης, εκφοβισμός από ομάδες συμφερόντων, από λόμπι. Και βλέπουμε επίσης εδώ ότι έχουμε και σωματικές επιθέσεις, σχεδόν 50%. Επίσης έχουμε παρενόχληση 13% ε, σεξουαλική παρενόχληση κατά γυναικών, κυρίως κατά γυναικών βεβαίως. 39% των απαντώντων μας είπαν ότι τους παρακολουθούσαν στοχευμένα, πολύ σημαντικό θέμα στις μέρες μας, και το οποίο αποτελεί απειλή κατά της προστασίας των πηγών. 76% λοιπόν των δημοσιογράφων αισθάνονται ότι δεν είναι επαρκώ προστατευμένοι προκειμένου. Και αυτό έχει επίδραση στην προστασία των πηγών. 48% των απαντώντων δήλωσαν ότι φοβούν ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν τι πηγές τους και ότι 25% αυτών είπαν ότι έχασαν τις πηγές τους λόγω αυτής τη κατάσταση. Επίση, απειλή χρήση δικαστικών μέσων, 23% δήλωσαν ότι συνελήφθησαν, ε, ήταν αντικείμενο διερεύνηση, ε, απειλήθηκαν με αγωγή ή ε, όντω ασκήθηκαν αγωγέ κατά αυτών των δημοσιογράφων και στι περισσότερε περιπτώσει ε, οι νόμοι που αξιοποιήθηκαν ήταν οι νόμοι περί δυσφήμισης. Έχουμε εκφράσει επανειλημμένω τη γνώμη μα περί αυτών, αλλά έγινε επίκληση και νόμων κατά τη τρομοκρατία, αντιτρομοκρατικών νόμων, προστασία τη δημοσία παρά την ανεπιθυμητή παρέμβαση πολύ μεγάλο ποσοστό, 35% των δημοσιογραφών ε, δήλωσαν ότι δεν έχουν επαρκή μηχανισμό καταγγελίας. Σε 40% είπαν ότι δεν ανέφεραν καν παρενόχληση στην ένωσή τους. Μετρήσαμε επίση ε, το θέμα του φόβου, δηλαδή την πιθανότητα άσκησης εκφοβισμού και στις, του φόβου εκ μέρους των δημοσιογράφων. Είναι μια μορφή βίας ή απειλή βίας. Και εδώ ψυχολογική βία, απειλές μέσω διαδικτύου κλπ. Όλα αυτά είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά. Πάνω από ένα τρίτο του Δήματος δήλωσαν ότι ανησυχούν σοβαρά για την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια φίλων και συγγενών και της οικογένειας. Μάλιστα αυτό είναι τόσο έντονο που 40% αυτών των ανθρώπων δήλωσαν ότι είχε επηρεαστεί η προσωπική τους ζωή. Η έρευνα βεβαίως έχει και άλλα συμπεράσματα. Εδώ σας παρουσιάζω μόνο τα κυριότερα. Πάντως αυτό σας δίνει μια ιδέα των ψυχικών επιπτώσεων και το στρες το οποίο προκαλείται. 37% των δημοσιογράφων είπαν ότι είχε επηρεαστεί και η δουλειά τους. Όλα αυτά βεβαίως ε, κατατείνουν προς την λογοκρισία. Εδώ τα αποτελέσματα είναι ζωφερά. 31% των απαντώντων δήλωσαν ότι είχαν τροποποιήσει ή αλλοιώσει ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, έγραφαν τα νέα. 19% είχαν προσαρμόσει το περιεχόμενο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εταιρείας, του εκδότη. 23% δεν δημοσίευσαν πληροφορίε που είχαν. Δεν έλαβα μας ζωφέρα. Κάναμε μια άλλη πολύ σημαντική ερώτηση. Η οποία έχει σχέση με το πώς αναπτύσσονται οι άνθρωποι μετά από κρούσματα βίας. Αυτό τους ισχυροποιεί. 36% λοιπόν είπαν ότι οι παρεμβάσεις αυτές ακριβώς τους έκαναν να προσκληθούν ακόμη περισσότερο στο ρεπορτάζ, στη δημοσιογραφία. Είπε μάλιστα κάποιος, έμαθα να εκτιμώ ε, αντιστρόφως τα αρνητικά σχόλια. Ήταν περιπτώσει που καταλάβαινα ότι είχα κάνει κάτι σωστό. Πολλοί λοιπόν δημοσιογράφοι συνεχίζουν ακόμα πιο ενδυναμωμένοι να υποστηρίζουν την αλήθεια. Επίσης ε, μελετήσαμε και γεωγραφικά την κατανομή αυτών των απειλών και εδώ θα σας πω για μερικά από τα αποτελέσματα, μερικά από τα πορίσματα σχετικά με την ε, διάδοση αυτών των κρουσμάτων. Επέλεξα αυτά που αφορούν κυρίως ε, τις χώρες μας αλλά και τις χώρες της περιοχής. Οι, φυσικές, οι σωματικές επιθέσεις ε, συμβαίνουν κυρίως στον Νότιο Κάφκασο και μετά στην Τουρκία. Συμβαίνουν όμως και σε άλλες περιοχές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μη ευρωπαϊκές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σε μη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερα προηγουμένω ότι έχουμε εδώ ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες και τα πάντα δεν είναι μόνο η συνήθιση, αν θέλετε, ύποπτη όπως λέμε. Συμβαίνουν όλα αυτά και σε χώρες που παραδοσιακά είναι δημοκρατικές και διαθέτουν ικανούς δημοκρατικούς θεσμούς. Και εκεί λοιπόν παρενοχλούνται οι δημοσιογράφοι. Σεξουαλική παρενόχληση, πρώτη Τουρκία και μετά ακολουθούν οι άλλες χώρες, αφορά κυρίως γυναίκες βεβαίως. Ψυχολογική βία, πολύ ψηλά σε όλες τις περιοχές, πάνω από 60% στην Τουρκία καταγγέλθηκαν τα περισσότερα κρούσματα στοχευμένης παρακολούθησης. Ε, Παρ' όλα αυτά, υψηλά ποσοστά είχαμε και σε όλες τις περιοχές και ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου, πρώτη Τουρκία και πάλι μετά η Νοτιοανατολική Ευρώπη και μετά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απειλή ε, αγωγών η συνήθις ε, επίκληση είναι του νόμου περί δυσφήμισης. Όπως προείπα και το είπε και η Ρενάτε νομίζω, η μελέτη καταλήγει σε συστάσεις. Καλή τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως αυτά τα οποία έχουν συνυπογράψει. Πρέπει να εφαρμόσουν λοιπόν στην πράξη τη συστάσεις του 2016 για την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων εργατών των μέσων ενημέρωσης να προλαμβάνουν τη βία, να προστατεύουν τους δημοσιογράφους, να προσάγουν και να μην αφήνουν τους τους παραβάτες και να ενημερώνουν γενικότερα τον πληθυσμό για την αξία της δημοσιογραφίας. Επίσης η μελέτη συνιστά στα κρατημέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να αξιοποιούν πλήρω την πλατφόρμα για την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε τον ε, Απρίλιο του 2015 και η οποία έχει σημειώσει, θα έλεγα, αρκετή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, θα ήθελα να μιλήσουμε για την συγκριτική, και μιλήσουμε για τη συγκριτική ανάλυση. Θα ήθελα να ακούσουμε τον καθηγητή Μπέρ Δέκα λεπτά πείτε μας τι έχετε εκεί. Γιατί κοιτάω το πρόγραμμα, όλοι έχουν την μελέτη. Πείτε μας τα βασικά. Πρόκειται για μια εξαιρετική μελέτη. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που έχει ζητήσει τον λόγο. Και έχουμε μέχρι τις 11. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη μελέτη αυτή και σας παρακαλώ πείτε μας τα κύρια σημεία. Σας ευχαριστώ. Τιμή μου να σας παρουσιάζω το έγγραφο αυτό το οποίο μας ζήτησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ το οποίο δημοσιεύτηκε από το Τμήμα Πολιτικής ε, Λίμπε. η έρευνα εξήχθη από τον καθηγητή Γιούρι Μπάιρ, Judith Μπάιρ, που κάθεται δίπλα μου και υπό την αιγίδα του τμήματος ε, δικαιοσύνης και ιστορικών του ΣΕΠΣ. Τώρα ο πλουραλισμός είναι ένα προαπαιτούμενο της ελευθερίας των ΜΜΕ και περιλαμβάνει όχι μόνο το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και τις διαφορετικές απόψεις στην κοινωνία. Αυτοί που χαράζουν πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εδώ και δεκαετίες εκφράσουν εκφράσει ανησυχίες για την σταδιακή περικοπή της ελευθερίας του πλουραλισμού των ΜΜΕ σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συνένεση για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό παρά το ότι σε όλα τα κράτη-μέλη οι επιχειρήσεις έχουν συνασπιστεί με τις πολιτικές δυνάμεις για να ασκήσουν πίεση στα ΜΜΕ τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές ε, και πολιτισμικές δυσκολίες ε, Η ψηφιοποίηση ανησύχησε πάρα πολύ τα ΜΜΕ. Η πρώτη μας υπόθεση όπως βλέπετε είναι πως όταν ε, συμπίπτουν οικονομικές και πολιτικές πιέσεις και υπάρχει εκμετάλλευση των νομικών παραθυρακίων υπάρχει συστημική παραβίαση τη ελευθερία των ΜΜΕ. Χωρί τα ΜΜΕ οι πολίτες δεν μπορούν να ελέγξουν ε, την κυβέρνηση ή να έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε για να ασκήσουν ε, τα πολιτικά τους δικαιώματα. Οπότε, το θέμα του πλουραλισμού θα συνδεθεί και συνδέεται με το ζήτημα της δημοκρατίας και θα αποτελέσει τμήμα του ελέγχου των πολιτικών ε, συναντικές πρόσφατες αλλαγές ε, στο ζήτημα της ε, δημοκρατίας σε κάποια κρατημέλη και η πρόσφατη αύξηση του λαϊκισμού και του εθνικισμού έχει δείξει ότι θα πρέπει να γίνει κάτι για να βελτιωθεί ο πλουραλισμός των ΜΜΕ. Τώρα, η υποχρέωση για πλουραλισμό προκύπτει από το δικαίωμα στην έκφραση. Το Δικαστήριο του Στρασβούργου έχει τονίσει πολλές φορές πως τα μέτρα των κρατών θα πρέπει να εγγυώνται αποτελεσματικό και ουσιαστικό πλουραλισμό. Αυτό έχει δύο πτυχές. Αφενός το κράτος μέλος δεν θα πρέπει να, το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει από την άλλη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει ποικιλομορφία απόψεων μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας και θεωρούμε ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς λέμε επιπλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να ρυθμίσει τα του πλουραλισμού στα μημία. Το επόμενο. Δεν υπάρχουν όμως αρμοδιότητες ε, παρόλα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν κάποιες άρρητες ε, αρμοδιότητες σε διάφορα επίπεδα του νομικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί, παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κάποιες συνέπειες όταν δεν γίνεται σεβαστό το άρθρο 11.2 της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μιλάει για πλουραλισμό των ΜΜΕ. Πέρα από αυτό υπάρχει και το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, παρά το ότι βεβαίως η χάρτα είναι κάπως περιορισμένη, η εφαρμογή της ισχύει πέρα από την ευρωπαϊκή του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και ήδη το δικαστήριο το έχει εφαρμόσει για τα κράτη-μέλη. Επίσης ε, το θέμα της επικότητας ε, της Ένωσης, η οποία περιέχεται σε ένα άρρητο κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες της ε, Ένωσης. Οι πολιτικές των κρατών μελών που εμποδίζουν τον πλουραλισμό των εμποδίζουν την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και υπηρεσιών. τέλο πρέπει να αναγνωρίσουμε πω όλοι οι μηχανισμοί επιβολή είναι εργαλεία κρίσης. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει ένας μόνιμος περιοδικός μηχανισμός παρακολούθησης των ΜΜΕ που θα βασίζεται σε αντικειμενικότητα και ισότητα για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους σε όλα τα κρατη Με λεπόμενη διαφάνεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε, στις 25 Οκτωβρίου 2016 να αποφάσισε να περάσει ένα ψήφισμα το οποίο ζητάει από την Κομισιόν να προχωρήσει νομοθετική πρωτοβουλία για έναν μηχανισμό για δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχει κάθε δυνατότητα να αποτελέσει την βάση μιας τακτικής αξιολόγησης δυνητικών κινδύνων στον πλουραλισμό των ΜΜΕ που προτείνουμε. Πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται σε κάθε κράτος μέλος από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών και εάν αξιολογείται ένα συγκεκριμένο σύστημα ότι εμποδίζει τον πλουραλισμό των ΜΜΕ, θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη συνεργασία με την κυβέρνηση για να βελτιωθεί σε βάθος πέντε ετίας ε, ο πλουραλισμός των ΜΜΕ. Τώρα, στην περίπτωση που αποκαλυφθεί ένας υψηλός κίνδυνος για τον πλουραλισμό ή αν η προηγούμενη πενταετής προσπάθεια έχει αποδειχθεί ανεπιτυχής, η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επιβολή είτε σύμφωνα με το άρθρο 258 της ε, συνθήκης είτε το άρθρο 7 είτε τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Για τις άλλες συστάσεις θα δώσω τώρα τον λόγο στην καθηγήτρια Μπάιερ. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την έρευνα, που κάναμε είχαμε το monitor για τον πλουραλισμό, το παρατηρητήριο για τον πλουραλισμό των ΜΜΕ 2014-2015 και βαστήκαμε και στην προηγούμενη έκθεση για τις περιορισμένες αρμοδιότητες της Ένωσης, αλλά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση μέσω συνεντεύξεων ε, ειδικών χωρών που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται σε κάθε χώρα. Θεώρησαμε ότι αυτό είναι αναγκαίο γιατί το θέμα αυτό εκφεύγει της ε, νομικής εποπτείας ε, και δεν είναι προφανές αυτό όταν το κοιτάει κανείς απ' έξω. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, το σπάσαμε σε μικρότερα υποερωτήματα, κυρίως να δούμε τον ρόλο του κράτους, την διαφάνεια και τις ε, παρεμβάσεις. Επιλέξαμε κάποια κράτη-μέλη όπου υποψιαστήκαμε ότι θα είχαμε κάποια αποτελέσματα. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ πέρα τα αποτελέσματα επιλέξαμε τις χώρες εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα τον κίνδυνο του πλουραλισμού από την πολιτική σκοπιά και την σκοπιά της ιδιοκτησίας. βέβαια δεν επηρεάζονται εξίσου όλα τα κράτη-μέλη, αλλά θεωρούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα κερδίσουν από τις συστάσεις αυτές όσον αφορά την διαφάνεια της ιδιοκτησίας, της ρύθμισης και εκπαιδευτικά προγράμματα. Επόμενη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, οι παράγοντες κινδύνου που βρήκαμε ήταν πρώτα απ' όλα η ιδιοκτησία που διαπλέκεται με κλάδους οι οποίοι αλλάσσονται με το δημόσιο και δεύτερον ή κρατικές διαφημίσεις που αποτελούν μια καλυμμένη μορφή επιδότησης. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα στην αγορά της Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Ελλάδας, ενώ στην Ιταλία και τη Γαλλία δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο και υπήρχε και ένα επίπεδο ρύθμισης της κατανομής της. Ε, βλέπουμε πως αυτά τα στοιχεία αποτελούν ένα άτυπο δίκτυο μεταξύ ΜΜΕ και πολιτικής και το επίπεδο της άτυπης επιρροής ε, θέτει αυτό το ζήτημα το οποίο πλέον από ποσοτικό γίνεται ποιοτικό ζήτημα πλουραλισμού και ελευθερίας. Επόμενη διαφάνεια βλέπουμε εδώ πέρα τι σημαίνει η λεγόμενη ήπια λογοκρισία χωρίς να υπάρχει άμεση λογοκρισία το κράτος μπορεί να επηρεάσει τα ΜΜΕ και από την πλευρά της χρηματοδότησης και του περιεχομένου μέσω διαφόρων κλάδων. Οι κλάδοι αυτή κατά κανόνα είναι η άμυνα ή οι δημόσιες μεταφορές, οι κατασκευές και επίσης ε, και η γη ε, περιλαμβάνεται στην Ουγγαρία γιατί λαμβάνει τεράστιε επιδοτήσει. Οπότε έχουμε άτομα τα οποία έχουν σχέση με την κυβέρνηση, στέλνουν ε, ευνοϊκά μηνύματα προς το ακροατήριό τους και μέσω αυτού του μηχανισμού έχουμε κάποιους πόρους οι οποίοι διοχετεύονται σε ιδιωτικές τσέπες και έτσι επηρεάζεται το περιεχόμενο από την ε, κυβέρνηση με τρόπο ήπιο αλλά ουσιαστικό. Έχουμε επίσης σχέση με πολιτική εξουσία σε που είναι άμεση σε Γαλλία, Ιταλία και Βουλγαρία και σε άλλες χώρες έμεση. Αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε ε, το τελευταίο έτος. Ε, δηλαδή διάφορα μήμοι ήταν στην ιδιοκτησία ατόμων που είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση και μπαίνουν τώρα στον κλάδο χωρίς να έχουν κάποια προηγούμενη σχέση με τα ΜΜΕ. Οπότε μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα τα οποία ουσιαστικά βάζει η κυβέρνηση να αγοράσουν κάποια ΜΜΕ, συχνά και με δημόσιο χρήμα ή με δημόσια χρηματοδότηση ή με δημόσια διαφήμιση. Επόμενη διαφάνεια. Οπότε τα συμπεράσματα είναι ότι αυτή η λογοκρισία δεν ε, επιβάλλεται μέσω νομοθεσίας περί λογοκρισίας, αλλά μέσω χρηματοδότησης και προσωπικών σχέσεων ιδιοκτητών. Δεν είναι προφανές δηλαδή για κάποιον εξωτερικό, χωρίς να γνωρίζει τους προσωπικούς δεσμούς που υπάρχουν στην κοινωνία, οπότε εύκολα αποκρύπτεται. Ε, Επίση υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη που εξετάσαμε, αλλά ιδιαίτερα στις νεότερες δημοκρατίες. Οι δεσμοί μεταξύ των ΜΜΕ και της κυβέρνησης είναι γνωστοί εδώ και δεκαετίες, αλλά στη συγκεκριμένη εποχή και χώρο ε, βλέπουμε ότι τα ΜΜΕ δεν ελέγχουν πλέον την εξουσία, δεν μιλάμε για λίγα ΜΜΕ, αλλά για όλα τα βασικά μέσα μιας χώρας. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι το σύνηθε σε μια Αφρικανική δικτατορία, αλλά αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω ε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παραβίαση δικαιωμάτων, αλλά όλο το σύστημα είναι διαστρεβλωμένο και με τη σειρά του επηρεάζει άλλα υποσυστήματα στη χώρα, κυρίω το πολιτικό σύστημα και την οικονομία όμω. Θεωρούμε ότι το δημοκρατικό αυτό έλλειμμα στο επίπεδο τη χώρα ε, πλέον ε, πλήττει το δημοκρατικό σύστημα, ειδικά τις εκλογές και τις ευρωεκλογές ε, λόγω της πολιτικής προπαγάνδας και των μηχανισμών αυτών. Επόμενη διαφάνεια. Ε, κοιτάξτε, ε, έχω δέκα ομιλητές λέει ο πρόεδρος. Ε, μα μου είχαν πει 15 λεπτά κύριε πρόεδρε. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, έχουμε τρεις σημαντικές εκθέσεις μετά από αυτό, μετά από αυτή την ακρόαση. Και ε, ήδη 10 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και πρέπει να απαντήσει και το πάνελ κάποτε. Όλα αυτά σε 20 λεπτά. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα γίνει. Οπότε σας παρακαλώ ε, σε να συντομεύετε. Ε, εντάξει, είναι μεγάλη δουλειά, αλλά θα γίνουν και ερωτήσεις. Ωραία, τελευταία διαφάνεια. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Όλοι έχουν την έκθεση. Καταλήξτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, οι συστάσεις. Ε, είχαμε τρεις, τρεις στόχους κατά νου. Πρώτον, οποιαδήποτε σύσταση που κάνουμε πρέπει να είναι βιώσιμη σε σχέση με τις υφιστάμενες αρμοδιότητες. Εστιάσαμε λοιπόν τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της Ένωσης όπως οι κρατικές ενισχύσεις, διαφάνεια κτλ. Δεύτερον, ότι θα πρέπει η νομοθεσία των κρατών μελών να παραμείνει. Και τρίτον, να είναι μικρές αλλαγές αυτές οι οποίες προτείνουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Και να γίνουν αποδεκτές βεβαίω. Αλλά θεωρούμε ότι εάν γίνει το πρώτο βήμα θα ξεκινήσει μια διαδικασία για να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές. Λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα τα βρείτε αυτά. Ναι, ναι, τα έχουν, τα έχουν, όλοι οι βουλευτές μπροστά τους. Οπότε, δείτε τις συστάσεις παρακαλώ, συνάδελφοι. Ε, που σας διακόπτω, είναι εξαιρετική η δουλειά σας. Απλά πρέπει να περάσουμε στους βουλευτές ε, που κάνουν τις ερωτήσεις, γιατί ε, δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε μετά τα επόμενα σημεία. Λοιπόν, περνάμε τώρα στους βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ε, δουλειά που κάνετε. Λοιπόν, αν θέλετε χρόνο να απαντήσετε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Κύριος Γιούρικ, παρακαλώ, σας παρακαλώ, δύο λεπτά ο καθένας. Αν έχετε ερωτήσεις για το πάνελ, παρακαλώ, απευθυνθείτε στα συγκεκριμένα άτομα που θέλετε. Λοιπόν, θα σας πω ποιοι συνάδελφοι ζήτησαν τον λόγο. Με τη σειρά που ζήτησαν θα δώσω τον λόγο. Γιούρικ. Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Κρίμα όμως που σε τούτη τη συζήτηση λησμονήσαμε κάποια στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά. Ας πούμε την δράση των κρατών. Ας πούμε, η πρόσφατη απόφαση ε, της ε, γαλλικής κυβέρνησης ε, που αφορά την απαγόρευση, ας πούμε, διακοπής κοίησης ή την απαγόρευση άσκησης ψυχολογικής βίας. Δηλαδή, υπάρχουν πολλών ειδών πιέσεις ε, στη διάρκεια ας πούμε του πολέμου του Βιετνάμ. Προφανώς ε, δεν μπορούσαν να γίνουν ε, πολλές συζητήσεις. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για κάποια θέματα για τα οποία έχει ασκηθεί πίεση. Τώρα, Εάν ε, πάρουμε τους ε, νόμους που αφορούν ε, την άμβλωση, Ξέρουμε ότι είναι πολλές οι δράσεις οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία του τύπου. Ας πούμε, χτες μιλήσαμε και προηγουμένως κιόλας για τις ψευδείς ειδήσει, fake news. Η απόφαση η οποία αφορά το ρομπέιτ είναι ένα είδος ψευδούς είδηση, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ελευθερία ε, του τύπου ε, και ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο επιλεκτική δικαιοσύνη. Ας πούμε, εάν μία φιλελεύθερη κυβέρνηση αρχίζει να παίρνει κάποια βήματα κατά της ελευθερίας του λόγου, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εάν μια συντηρητική κυβέρνηση ε, αρχίζει να κάνει το ίδιο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Mr. Boney, please. Thank you. Boney. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πρώην αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες ε, για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν και οι οποίες ε, είναι πραγματικά ιδιαίτερα πλούσιες και μας δείχνουν και φωτίζουν πολλές πτυχές του θέματος. Οι ψευδείς ειδήσει, η πίεση για λογοκρισία και αυτολογοκρισία είναι θέματα πολύ σημαντικά. Εγώ είμαι Πολωνός και αυτά όλα, αυτούς όλους τους περιορισμούς ε, της ελευθερίας των μέσων ε, τις αισθάνομαι πολύ πιο έντονα. Τώρα Μιλάμε για ε, μεταφορά των πληροφοριών που πρέπει να ξεχωριστεί από την προπαγάνδα. Θα πρέπει ε, ε, επίσης να πούμε ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ε, και το θέμα της έλλειψης ουδετερότητας, της μείωσης της ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου στην ε, Ευρώπη υπάρχουν, υφίστανται ήδη οι μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε τέτοιου είδους παρεμβολές, τέτοιου είδους παρεμβάσεις από πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις κλπ. να ε, ε, μην υφίστανται ή να μειωθούν πολύ. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η υπερσυγκέντρωση των μέσων ε, ενημέρωσης. Θα πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση, αλλά μερικές φορές αυτή ακριβώς ε, η προσπάθεια αποκέντρωσης ε, καταστρέφει κάποια μέσα ενημέρωσης από ε, ευρωπαϊκής πλευράς θα πρέπει να τα δούμε όλα τα θέματα αυτά ε, κάτω από ένα νέο φως και κάτω από ένα νέο πρίσμα βεβαίως γνωρίζω ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο έγινε λόγος επίσης ε, για, τον, για την εργασία των δημοσιογράφων είναι πολύ σημαντική η εργασία των δημοσιογράφων και το έργο τους υπέρ της ελευθερίας ευχαριστώ πολύ Άννα Γκόμες Ευχαριστώ για την διοργάνωση της ακρόασης. Εγώ θέλω να τονίσω πόσο εμένα ως Πορτογαλίδα μου έκανε αίσθηση η αναφορά στην υπερσυγκέντρωση. Η Κομισιόν δεν τα λεφτά στη χώρα μου. Η πρώτη κίνηση έγινε από πλούσιες οικογένειες από την Αγγόλα Δεν ήταν ότι έβγαζαν λεφτά, αλλά ήθελαν να ελέγξουν τις εξελίξεις ε, στην Πορτογαλία. Ήθελαν να ελέγξουν τη ροή των ειδήσεων. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα τα μέσα στην Πορτογαλία κάνουν φανταστική δουλειά. Τα μέσα, αυτή τη στιγμή είδατε τι έγινε με τα Panama Papers. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος για τις μεταφορές σε εξωχωρές εταιρείε επί τρόικα 10 δισεκατομμύρια έφυγαν από την Πορτογαλία και πήγαν σε ξεχωρίες εταιρείε. Τι γίνεται με την διαφάνεια, με τι πρόσφατε φωτιέ, με την κλοπή πολεμικού υλικού στην Πορτογαλία. Σε όλα αυτά τα μέσα βοήθησαν πάρα πολύ. Με προσωπικό κόστο, σε πολλέ περιπτώσει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και σε εμά υποφέρουν οι δημοσιογράφοι και δέχονται απειλέ, όπω παντού, εκφοβισμό, εκφοβισμό μέσω διαδικτύου, τη σωματική του ακεραιότητα κλπ την Ουγγαρία και την Τουρκία. Τώρα η κατάσταση είναι ιδιαίτερω ανησυχητική, όπω είπατε και εσεί. Έχω μία ερώτηση. Έχουμε και το Euronews, όπω ξέρουμε. Έχουμε το Euro μπροστά. Υποτίθεται ότι εκεί υπάρχει πολλή ελευθερία, αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητο ρεπορτάζ κλπ. Όμως, ακούσαμε ξαφνικά ότι υπάρχουν προβλήματα στο Euronews λόγω ελέγχου από ξένα κεφάλαια. Δεν είναι μόνο το Sky και Fox. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε πολιτική θέση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να συζητάμε για δυσφημίσεις, για απειλές κλπ. Ε, ε, Θυμάρα των οποίων έχω υπάρξει και εγώ. Και το Euronews με απείλησε με αγωγή για δυσφήμιση κατά του Euronews. Επειδή είπα ακριβώ αυτά που λέω τώρα, δεν προχώρησε. Λοιπόν, μήπως είναι καιρό να το δει πολιτικά η Κομισιόν επιτέλου το θέμα. Να κάνει τη δουλειά της, την ευρωπαϊκή της δουλειά βάσει των στόχων της συνθήκης υπέρ της δημοκρατίας και όχι για να μην το δει μόνο ως οικονομικό θέμα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Η πολυφωνία είναι κρίσιμη σημασία, εννοείται, για το κράτος δικαίου, την φιλελεύθερη δημοκρατία κλπ. Όμως, έχω και κάποιες ε, επικρίσεις και κάποια επιμάχα θέματα. Πρώτον, αναφέρθηκε σε διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να θέλω φλούμε. Πρέπει να είναι σαφές. Ε, μπορεί να έχουμε τα θέματα μας με την Τουρκία και το Μοντενέγρο, αλλά δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον, η Πολωνία και η Ουγγαρία, συστηματικά, συστηματικά ταπεινώνουν την ελευθερία του τύπου και των μέσων. Δεν είναι σαφές ότι η δημοκρατία χρειάζεται πάντοτε ανεξάρτητα πολυφωνικά μέσα. Και αυτό αφορά εμάς. Δεν χρειάζεται να πάμε παρέξω. Αυτά σημαίνουν στο σπίτι μα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Τουρκία. Και κύριε Μπέρμαν, Αναφέρατε την δύσκολη κατάσταση των εντύπων μέσων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολύ σημαντικό θέμα. Δείτε τι γίνεται με τα τοπικά μέσα στην Ουγγαρία ή στην Πολωνία, όπως προείπα, που αποτελούν πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών, πολιτικών και άλλων πληροφοριών για την περιοχή. Πρέπει λοιπόν να το πούμε αυτό φωναχτά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, τα ψευδονέα, ψευδοειδήσεις που χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα είναι η επίσημη πολιτική των δύο κυβερνήσεων, της Ουγγρικής και της Πολωνικής κυβέρνησης. Μην υπεργενικεύουμε. Εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα. Και γι' αυτό είναι αδερήτη ανάγκη να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητές μας στον τομέα ακριβώς της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων. Βασιλικιάκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που ε, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Εξ αρχής θα πω ότι ναι, όντως είναι αλήθεια ότι δεν θα πρέπει ε, να ξεχάσουμε, να απαρνηθούμε τις αρχές και τις ελευθερίες τις δημοκρατικές. Γιατί πραγματικά εντός της ελευθερίας θα πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί και η ελευθερία και η πολυφωνία του τύπου. Ωστόσο θα υποβάλω και ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι οι ψευδείς ειδήσει αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία. Ε, είναι ε, ακριβώς ένα πρόβλημα το οποίο αφορά και στο, ε, στο θέμα της μετάβασης στην ψηφιοποιημένη εποχή. Οι ψευδείς ειδήσει τελικά κατακλείζουν το δίκτυο το οποίο έχει γίνει ένα no man's land. Ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε, να κάνει οτιδήποτε και ταυτόχρονα να έχει έναν μεγάλο αντίκτυπο. Απειλεί λοιπόν στη δημοκρατία εξού και η ευθύνη της Ευρώπης ε, και των θεσμών της ε, να βάλει κανόνες. Ε, οι κανόνες θα πρέπει να είναι πολιτιστικοί αλλά οπωσδήποτε και νομοθετικοί. Ερώτηση, ποια είναι η κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, κάτω από την οποία κόκκινη γραμμή δεν μπορούμε να κατεβούμε, ενδεχομένως μαζί μέσω αυτού του διαλόγου θα μπορούσαμε να καθορίσουμε αυτή την κόκκινη γραμμή. Γιατί κατά την άποψή μου αυτός ο χώρος που δεν ανοίξει κανέναν θα μπορούσε να είναι και ο χώρο με, εντός του οποίου ο καθένα μα μπορεί να φανεί ισχυρό. Ευχαριστώ η κυρία ε, Καρπίνη. prezentat experții în studiile pe care le-am uh, văzut, lucruri interesante pentru fiecare dintre noi. Adresez o întrebare. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Οι ψευδείς ε, ειδήσει οπωσδήποτε είναι κάτι ε, που αφορά όλους, αφορά όλους τους ανθρώπους και ε, μακροπρόθεσμα αφορά και επηρεάζει και την ποιότητα της δημοκρατίας. Μιλάμε για άλλη δημοσιογραφία, για δημοσιογραφία άλλης ποιότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει ε, την δημοκρατικότητα των μέσων ενημέρωσης. Δεν θεωρείτε ότι η δημοσιογραφία κακής ποιότητος και οι ψευδείς ειδήσει σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, γράφονται από δημοσιογράφους οι οποίοι πληρώνονται για να ε, διαδώσουν τις ψευδείς ειδήσει, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει και μία ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη, την υπευθυνότητα και την ελευθερία. Θα πρέπει ο καθένας μας να είναι υπεύθυνος. Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι εξαιρετικοί οι οποίοι αποκαλύπτουν τρομερά σκάνδαλα, αλλά υπάρχουν και, και αυτοί μάλιστα ε, υφίστανται απειλές, εκτονούς κτλ. ενώ υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι γράφουν ε, άρθρα κακής ποιότητας και που τους αφήνουν όλους ε, ήσυχους. Thank you. Sophie Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές και την Μπάρμπαρα Σπινέλη, την εισηγήτρια. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην συμφωνία ε, στην ελευθερία και τον πλουραλισμό του ΜΜΕ, αλλά όταν ε, μιλάμε για πρακτική εφαρμογή είναι λίγο δύσκολο. Και γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί τα ΜΜΕ δεν αφορούν πλέον μόνο τη μουσιογραφία, αλλά έχουν περάσει στα κοινωνικά μέσα και εκεί πέρα έχουμε διάφορα παράδοξα γιατί οι ψευδείς ειδήσει κατά κάποιον τρόπο είναι επίσης μέρος της ελευθερίας έκφρασης και του πλουραλισμού. Και ποια είναι η πηγή των ψευδών ειδήσεων, αν είναι ένας δημοσιογράφος, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για διοντολογία της δημοσιογραφίας. Αλλά είναι κάποιος άλλος ή και πολιτική. Υπάρχουν και πολιτικοί και... και ηγέτες του δυτικού κόσμου που λένε μπούρδε. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για περιορισμό ψευδών ειδήσεων. Ε, ο Τάις Μπέρμαν έχει δίκιο. Πρέπει απλά να το αντιμετωπίσουμε με το να λέμε την αλήθεια. Συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπε ο Τάις Μπέρμαν για την ελευθερία των δημοσιογράφων που απειλείται από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, αλλά πέφτει όταν μη ακουόντων. Και δυστυχώς αυτές τις μέρες θα περάσει τη σχετική νομοθεσία η Ολλανδική Βουλή, κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ελευθερία της δημοσιογραφίας και των πηγών των δημοσιογράφων. Αυτό είναι πολύ άσχημη εξέλιξη. Κάποιος ανέφερε τους νόμους περί φήμησης που αποσύρονται, αλλά οι νόμοι περί βλασφημίας υφίστανται και έχουν εισαχθεί και νέοι σε κάποια κράτη-μέλη και εφαρμόζονται. Και αυτό πρέπει να δούμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, για τη για τα περισσότερα δημόσια ΜΜΕ, τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα δημόσια ΜΜΕ. Ακούγεται καλή ιδέα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο εδώ πέρα πολιτική παρέμβαση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι απόψει σα μετά. Για την ιδιοκτησία των ΜΜΕ και την ε, συγκέντρωσή τους που ανέφερε ο κ. καθηγητής. Έχετε αξιολογήσει την υπερσυγκέντρωση μόνο ανά κράτο ή εξετάσατε και την διασυνοριακή ιδιοκτησία και το τι σημαίνει αυτό για τον πλουραλισμό. Και δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Κάτι το οποίο νομίζω έθιξε και ένας προηγούμενος ομιλητής. Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι επίσης πρέπει να κάνουν αυτή τη συζήτηση αλλά και τη συζήτηση για την δημοσιογραφική ιδεοντολογία, γιατί θυμόμαστε σκάνδαλα όπως το News of the World. Και βεβαίω θα μιλάμε για την υπερσυγκέντρωση των ΜΜΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, δεν γράφουν οι ιδιοκτήτες τα άρθρα, είναι οι δημοσιογράφοι. Οπότε και αυτοί πρέπει λίγο να α, το δουν το πράγμα. Και μια, μια τελευταία παρατήρηση. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο η παρακολούθηση του προελισμού των ΜΜΕ πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός, όπως είχαμε συμφωνήσει κατ' επανάληψη στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να αποτελέσει ένα τμήμα τη γενικότερη αυτή έκθεσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί του χρόνου δεν θα πρέπει να έχουμε μια χωριστή έκθεση για τα ΜΜΕ, αλλά μια ενία. Ε, Σόφι, σε παρακαλώ, συντόμευε. Κίνγκα Γκάλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές ε, που μοιράστηκαν τις διαφορές ιδέες τους μαζί μας. Στην ακρόαση αυτή. Κοιτάξτε. Ναι, κάτι δεν άκουσα εγώ ε, που θα ήθελα να ακούσω. Δηλαδή η διάδοση ψευδών ειδήσεων είναι ένα πρόβλημα και όπως είπαν κάποιοι υπάρχει γενικότερη πτώση της ποιότητας ε, της δημοσιογραφίας και του επαγγελματισμού. Η έκθεση Λίμπε τώρα παρήγγειλε μία έκθεση και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ. Και πρέπει να πω ότι κάποια τμήματα αυτής της έκθεσης αφορούν την Ουγγαρία. Εγώ είμαι Ουγγαρέζα και αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για θεωρίες συνωμοσία που υπάρχουν και Πραγματικά ε, δεν ξέρω ποιε είναι οι ψευδεί ειδήσει. Ε, δηλαδή μιλάμε για προδοσίες, ε, συνωμοσίε, η έκθεση αυτή παριστάνει την επαγγελματική αλλά περισσότερο αρμόζει σε ένα ταμπλόιντ. Απορρίπτω την ιδέα ότι είναι επαγγελματική αυτή η έκθεση. Αναπαράγει ιστορίες τελείως αστήρικτες, αναλυθείς ή στην καλύτερη περίπτωση βασίζονται σε πολύ υποκειμενικά στοιχεία ή σχόλια στο facebook ή κάτι περίεργα άρθρα στην Ουγγαρία και δεν θα έπρεπε τώρα να έχουν θέση αυτά σε οποιαδήποτε έρευνα του Κοινοβουλίου. Ο πλουραλισμός των ΜΜΕ λοιπόν δεν έχει περισσότερα προβλήματα στην Ουγγαρία από ό,τι σε άλλες χώρες. Γιατί βλέπουμε ότι κάποια από την κριτική από τις ε, ε περίεργες αυτές πηγές ε, δημοσιεύεται, ε, βρίσκει ε, λόγο και στην έκθεσή σας, οπότε βλέπω το ζήτημα της ε, ελευθερίας που υπάρχει. Λοιπόν, εμείς ζητήσαμε αυτήν την έκθεση και δεν ερωτήθηκαν ε, διάφοροι, διάφορα θεσμικά όργανα για το αν ισχύει αυτή η έκθεση, αλλά θα βασιστούν σε αυτήν και λυπούμε για όσους θα λάβουν αποφάσεις ε, επί τη βάση τελείως υποκειμενικών πληροφοριών του πληροφοριών του είδους που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Παραδείγματος χάρη ε, την ιδέα, η ιδέα ότι το άρθρο 7 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ε, σύμφωνα με ε, το άρθρο 285 έχουν εντύπωση ότι έχετε, είχατε καταλήξει τα συμπεράσματα εκ των προτέρων και έγινε κατόπιν εντολής. Κύριος Μέλλον. Ο τύπος είναι η ελευθερία. Τύπος σημαίνει ελευθερία. Και σήμερα και χθες και αύριο. Τι βλέπουμε όμως. Τα κόμματα εκμεταλλεύονται τη δημοσιογραφία. Συμβαίνει συνεχώς, συμβαίνει παντού. Το πολιτικό κίνητρο υπάρχει. Και το φαινόμενο είναι πολύ σοβαρό. Σε Κάποιες χώρες, οι δημοσιογράφοι τροποποιούν το μήνυμα, είναι προφανές, σε αρτήση των πολιτικών συμφερόντων. Δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, πολύ απλά. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πολιτικοί έχουν στη διέθεσή τους πλέον ένα εξαιρετικό εργαλείο για να παίρνουν πολιτικά μηνύματα χωρίς ε, να παίρνουν μέσω του τύπου να μια απειλή για τον τύπο στο μέλλον. Ποια είναι η σχέση λοιπόν μεταξύ δημοσιογράφων και μέσων, των νέων μέσων αν θέλετε και πώς βλέπουν οι δημοσιογράφοι το ρόλο τους ε, εν ώψη και του ρόλου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαδερματίζουν όλο και ισχυρότερο ρόλο. Κάτσε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ε, καλεσμένους μας ε, που ε, ε, μας παρουσίασαν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα εξαντλητικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως την συνάδελφο Σπινέλη με την οποία θα συνεργαστούμε μαζί με τους Κιώδης επί της εκθέσεως. Ήδη από την αρχή ο καθηγητής κ. Πάρκου ανέφερε ότι νομοθετικά στην Ευρώπη η κατάσταση είναι καλή αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι διαφορετικής ένταση ο καθένας. Ε, η κυρία Σρέντερ μα είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό περιβάλλον όπου θα προστατεύεται το δημοσιογραφικό επάγγελμα απέναντι σε προβλήματα, απειλέ κτλ. Και ότι υπάρχει σχετική σύσταση και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναρωτιέμαι για αρκεί αυτό ε, για να διασφαλιστεί η προστασία των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας ή χρειάζεται και κάτι άλλο. Προλαλήσαντες ανέφεραν ψευδείς Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει για τις ψευδείς ειδήσει να πάρουμε θέση και να πάρουμε και μέτρα, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία έκφραση και την ελευθεροτυπία από τη μία ε, και ε, στην ανάγκη να μειωθούν οι δημοσιευμένες ε, ψευδείς ειδήσει. Επίσης, το θέμα της πρόσβασης των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Οι γυναίκες δυστυχώς υφίστανται περισσότερο εκφοβισμό, περισσότερες και εδώ τι μπορούμε να κάνουμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να παρεύουμε για το θέμα αυτό, το οποίο μου φαίνεται και αυτό εξαιρετικά σημαντικό. Και τέλος, το ε, έθιξε και η, κυρία Σπινέλη. Ε, το θέμα της advocacy νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε θέση. Ε, και επ' αυτού θα ήθελα επίσης να, να γνωρίζω την άποψη των εισηγητών. Um, I just had one last... Πολύ ωραία. Και μια γρήγορη ερώτηση προ την κυρία Είναι ερώτηση της κυρία Σιντεβέλτ σχετικά με την κατάσταση των μέσων. Ανέφερε την υπερσυγκέντρωση της ιδιοκτησία και είπε ότι θα μπορούσε να ενορχιστρωθεί μια μαζική επίθεση κατά ενός ή άλλου κόμματος μέσω και των ιστοτόπων μαζικές ε, επιθέσεις κατά ας πούμε, γυναικών πολιτικών. Οι ιδιοκτήτες πλέον μπορούν να ενορχιστρώσουν, όπως είπα, τεράστιες μαζικές επιθέσεις εν ώψη και εκλογών κατά πολιτικών, κατά γυναικών, κατά χρώμων, κατά ανθρώπων που υποστηρίζουν συγκεκριμένες απόψεις, προσπαθώντας λοιπόν να τους σταματήσουν, να τους κάνουν να σιωπήσουν με εκστρατείες, με λασπολογία κλπ. Ποιο είναι ο ψυχολογικός αντίκτυπο όλων αυτών. Το βλέπουμε κυρίως στι ΗΠΑ. Δεν είναι αλήθεια ότι ακόμα και καλοί δημοσιογράφοι απειλούμενοι κάνουν συμβασμούς. Υπάρχουν παντού καλοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν είναι σε κίνδυνο να απειλούνται από τους ιδιοκτήτες. να ξεκινήσουμε δεξιόν μου και υπάρχουν. Θέλετε να πείτε δύο λόγια για τα βασικά πράγματα που ακούσαμε. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε στα πάντα. Τα βασικά μόνο. Δύο βασικά μηνύματα. Δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ. Είστε σύντομοι. Θίξτε μόνο αυτά τα οποία θεωρείτε εσείς πιο σημαντικά. Παρακαλώ. Δύο-τρία λεπτά. Για να δώσω το λόγο και στους άλλους παρευρισκομένους. και για να κλείσουμε. Πρόεδρε. Έχουμε αυτή την ομάδα για τις ψευδοειδήσεις, έχουμε και ένα σεμινάριο αύριο. Είναι και στο κέντρο της δουλειάς μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για τις ψευδοειδήσεις είναι να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους από, την, από τις πολιτικές και οικονομικές εξωτερικές παρεμβάσεις. τα βασικά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά ανεξαρτησία στο γράψιμο, στη σύνταξη. Να δίνουν στον κόσμο την αλήθεια και να μην είναι υποκείμενοι σε εξωτερικές παρεμβάσεις. Και μετά, βεβαίω, έχουμε τα άλλα θέματα, έχουμε το διαδίκτυο, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα νέα ειδήσει στο διαδίκτυο. Θέλει εις βάθος μελέτη το πράγμα. Θα ξεκινήσουμε ένα τέτοιο, τέτοια μελέτη στο Ινστιτούτο μα. όμως το βασικό είναι, η αρχή των πάντων είναι να προστατεύσουμε του δημοσιογράφου, την ανεξαρτησία των μέσων. Να προστατεύσουμε τα μέσα από την υπερσυγκέντρωση τη ιδιοκτησία στα χέρια ολίγων. Και δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τη διασυνοριακή συγκέντρωση, όσο για τη συγκέντρωση εντό μια συγκεκριμένη χώρα ή τη συγκέντρωση διαφορετικών μέσων στα χέρια ενό. Η τη συγκεντρωση διαφορετικων μεσων στα χερια ενο η διασυνοριακη συγκέντρωση μπορεί να γίνει πρόβλημα. Αργότερα όμως είναι ένας ε, τρόπος κάποιοι να ελέγξουν κάτι και μπορούμε να κάνουμε κάτι νομίζω προς το παρόν για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε από το... ενώψη μελλοντικών εξελίξεων. Ε, γυναίκες τώρα και μειονότητες, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Εδώ θέλει περαιτέρω μελέτη. Και πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και κάτι πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Και κάτι άλλο που υπόθηκε βεβαίως, ναι, Τουρκία και Μαυροβούνιο συμφωνεί. Και μάλιστα κυρίως το Μαυροβούνιο σε κάποιους τομεί. Δεν πάνε και πολύ καλά, αλλά και χώρε ευρωπαϊκέ, με κάτι μέλη. Μην νομίζετε ότι δεν είναι στο, στο σκοπευτρό μας. Γι' αυτούς τους λόγους πάντως, ε, και επειδή έχουμε ένα κεφάλαιο στις υποψήφιες χώρες που αφορά τα μέσα, να κάνουμε τέτοιε αξιολογήσει για τα ήδη κράτη-μέλη και όχι μόνο για αυτού που θέλουν να γίνουν μέλη. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομο, ευχαριστώ πολύ και πάρκο και πέρμεν. Κλοντ. Κλοντ, ευχαριστώ και για τις ε, παρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις σας για την Γαλλία. Κύριε Γιώργο, μια βδομάδα μετά την κηδεία της Σιμών Βέιλ, που ήταν ηρωίδα στην Γαλλία, ε, οφείλω να σας απαντήσω. Η ελευθερία των γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα τους ε, έχει περάσει το γαλλικό νόμο και υπάρχει συζήτηση στην ε, γαλλική κοινωνία, βεβαίως ε, ο νόμος υπάρχει. Η κόκκινη γραμμή για τις ψευδείς ειδήσει είναι ακριβώς η λογοκρισία. Γιατί η λογοκρισία οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε περισσότερη λογοκρισία. Και θα βλάψει την κοινωνία και τα άτομα. Είναι πολύ απλή η γραμμή λοιπόν. Όχι λογοκρισία. Αλλά να αποκαλύψουμε την παραπληροφόρηση αυτό σχετίζεται με την αυτορύθμιση και την ε, επαγγελματική ιδεοντολογία των δημοσιογράφων που πρέπει να είναι σαφής για τους ιδιοκτήτες των μέσων, για τις πολιτικές τους επιλογές, έτσι ώστε ένα πολιτικό σχόλιο ενός δημοσιογράφου στην εφημερίδα του ΙΤΙΣ να έχει μια ξεκάθαρη πηγή και ο κάθε πολίτης μετά θα κρίνει αν θα το δεχτεί ή όχι. Συχνά οι εφημερίδες δεν είναι ρητή. ρητές, για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Για τα συμφέροντα. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουν οι πολιτικοί όμως. Οι, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να το κάνουν οι πολιτικοί, έτσι θα περιοριστεί η ελευθερία της έκφρασης και των μημιών. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε δηλαδή ακριβώς. Η βλασιμία. Πράγματι, Σοφίνετφελντ, υπάρχει στην ομοθεσία πολλών χωρών ακόμα. Καλύτερο θα ήταν βεβαίω να φύγει, αλλά το ίδιο ισχύει και για την δυσφήμιση. Προσφάτως ένας Έλληνας μουσιογράφος ε, υπέστη ε, ένα ε, πρόστιμο 1.500 ευρώ επειδή περιέγραψε ένα μέλος Χρυσής Αυγής ως ε, νεοναζί και αυτό έκρινε το δικαστήριο ότι ήταν δυσφήμιση. Κάτι το οποίο βεβαίω το ότι το θεώρησε δυσφημιστικό είναι ε, θετικό από την άλλη. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε και σύντομοι. Λοιπόν, ένα σόρτα. Ναι, θα συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσαντες για τις ψευδείς ειδήσει. Ναι, όπως είπα, η συζήτηση είναι πολιτική, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στον δημοσιογραφό και στη δημοσιογραφία. Πάντα υπήρχαν ψευδείς ε, ειδήσει και το θέμα είναι τώρα η ταχύτητα και το πόσο γρήγορα διαδίδονται και τα κοινωνικά μέσα, ότι ο κόσμος απευθύνεται απευθείας μέσω ε, του Facebook και παρακάμπτει τους δημοσιογράφους επενδύσουμε τώρα στη δημοσιογραφία. Μου θυμίζει τη συζήτηση για τη δημοσία χρηματοδότηση. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά μοντέλα. Δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο. Σαφές επίσης το ότι υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια. Το ένα είναι να επενδύσουμε στα δημόσια μήμιε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει βεβαίως ε, το πρόβλημα το οικονομικό αλλά πρέπει να υπάρχει και πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία. Καλό θα ήταν επίσης να υπάρχει και χρηματοδότηση για διάφορα ερευνητικά έργα. Το είδαμε και πριν από το Panama Papers. Έχουμε δει την ε, σημασία που έχει αυτό σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και οι πλατφόρμες των πολιτών θα είναι χρήσιμες, αλλά νομίζω ότι είμαστε στην αρχή ακόμα. Όταν μιλάμε τώρα για αυτό το οποίο είπατε και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα που έχουμε με την υπερσυγκέντρωση των ΜΜΕ, τους πολιτικούς λοιπά. Θα συμφωνήσω και εγώ, αυτορύθμιση, ιδεοντολογία, αλλά υπάρχει και η επισφάλεια των δημοσιογράφων. Όταν βγάζουν λιγότερο από 10 ευρώ ε, αναρεπορτάζ, ε, δεν υπάρχει ποιότητα. Είναι μια συνολική προσέγγιση λοιπόν αυτή που πρέπει να υπάρξει. Και πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάτε τώρα περνάμε στον καθηγητή, στην καθηγήτρια Κλάρκ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί υπόθηκαν πολλά. Νομίζω ότι το θέμα της λογοκρισίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το, νομίζω ότι θα πρέπει σαφώς να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εντός του οποίου μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι δημοσιογράφοι και επομένως ένα περιβάλλον χωρίς φόβο, χωρίς εκφοβισμό, ανεξάρτητο. Ε, ε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάποιους ε, νόμους που αφορούν την επιτήρηση και την παρακολούθηση ε, που είναι πάρα πολύ προβληματικοί όσον αφορά την προστασία των πηγών. Αυτά. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαίρετη η συμβολή όλων σας. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγο αν πούμε ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο, αλλά ε, βεβαίως το σημαντικό ε, είναι και λαμβάνοντα υπόψη τα όσα έχουν λάβει χώρα φέτος, να πούμε ότι απλώς υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ε, αφορούν συγκεκριμένε χώρες, αλλά ότι το θέμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης είναι ένα γενικευμένο ζήτημα το οποίο ξεπερνάει τις μεμονωμένε χώρες. Ε, θα ήθελα να δώσω τον τελευταίο λόγο για τα συμπεράσματά της στην ε, εισηγήτρια. Όπως ξεκίνησε έτσι θα κλείσει η συζήτηση ε, με την εισηγήτρια και τη ζητώ να κλείσει και την ακρόαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Σπινέλη. Σας ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πολύ σύντομα κάποια στοιχεία. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λειτουργεί καλά στα κριτήρια και στους δείκτες που αφορούν την ελευθερία του τύπου. Εάν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ε, εμφανίζεται μεταξύ των χωρών ε, που ε, σέβονται περισσότερο από άλλους την ανεξαρτησία του τύπου. Εάν υπάρχει μια χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του τύπου ε, παρήγαγε ψευδείς ειδήσει σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο του Brexit ήταν ακριβώς το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως θα πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε λίγο τους δείκτες μας. Δεύτερο προς απάντηση σε αυτά που είπε η Μάριλιν Κλάρκ. Να πω ότι δεν παρηγοριέμαι και πολύ, δεν είναι μεγάλη παρηγοριά ε, όταν ε, λέμε ότι το τραύμα ενός ε, δικαίου που δεν έχει ληφθεί υπόψη μπορεί να ξεπεραστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει χρήσιμο κακό, δεν υπάρχει τραύμα το οποίο έχει λόγο ύπαρξης. Επίσης, κόκκινες γραμμές ε, και νομοθετικές ρυθμίσεις. Ε, πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον δόκτωρα Μπέρμαν. Αυτό που πρέπει ε, πάντα να προτιμούμε είναι η αυτορύθμιση από πλευράς του κόσμου της πληροφορίας και των δημοσιογράφων. Οι κρατικές αποφάσεις είναι πάντα επικίνδυνες. Τελευταίο, έχουμε δύο καλά άρθρα τα οποία υπεραμείνονται της ελευθερίας του τύπου. Το άρθρο 10 ε, της ε, ε, Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου γίνεται αναφορά όχι μονάχα για το δικαίωμα του δημοσιογράφου να πληροφορήσει, αλλά και αναφέρεται και στο δικαίωμα του πολίτη να πληροφορηθεί. Υπάρχει δηλαδή το εξειδικευμένο δικαίωμα του αναγνώστη ή του θεατή που βλέπει ε, τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, εξίσου σημαντικό το άρθρο 11 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνει ένα στοιχείο που δεν αναφέρεται στη σύμβαση. Αναφέρεται λοιπόν στην πολυφωνία και όχι μόνο στην ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλου και ευελπιστώ ότι θα παραμείνουμε σε επαφή και του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ πρόεδρο ευχαριστώ πολύ ε, Μπάρμπαρα. Ε, ξέρω ότι όλα αυτά αυτά θα συμπεριληφθούν στην έκθεσή σου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ε, πραγματικά ήταν εξαίρετη η τον αλλο τροπο πραγματικα ηταν εξαιρετη η ακροαση Ε, σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ ε, για αυτήν την ακρόαση όλους σας. Θα προχωρήσουμε τώρα σας ευχαριστώ πολύ, ε, όπως είπα και προηγουμένως όλους όσοι συμμετείχατε ε, στην ακρόαση. Θα συνεχίσουμε τώρα με, την, ε, με τις εργασίες.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 And we move to point 13, Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως που αφορά πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων της ένταξης των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πολέμηση του αντιαθηγανισμού. Πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα, λέει ο Λοιπόν, το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ε, Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα μελετούμε το ε, ευρωπαϊκό πλαίσιο ένταξης των Ρωμά που ξεκίνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που προβλέπει η προστασία και επιτήρηση και στα κράτη-μέλη. Πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα, γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια, ε, η οποία είναι εισηγήτρια για ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με θέμα πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων της ένταξης ε, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί μπορούμε να ακούσουμε την παρουσίαση του προσχεδίου έκθεσης της κυρίας Σοράγια Πόστ, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο.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 Ε, θα ήθελα πρώτα να σας πω ότι οι προηγούμενοι μήνες, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν πάρα πολύ καλή για μένα. Η κατάσταση όσον αφορά τους Ρωμά ε, ήταν και εξακολουθεί να ε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για τους Ρωμά. Τις περισσότερες φορές όμως πρέπει να αγωνιστούμε ιδιαίτερα έτσι ώστε να έχουμε έστω και μια μικρή προσοχή όσον αφορά τα θέματα. Η προσφυγική λεγόμενη κρίση είναι αυτή η οποία τελικά παίρνει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά το ενδιαφέρον του κοινού και ε, των κρατών. Ε, και επομένως ε, ο αντιεθνικανισμός μπορεί να έχει πάρα πολλά πρόσωπα και να βρίσκεται σε πολλά επίπεδα. Μπορεί δεν να εκδηλώνεται ε, ε, με πολλούς τρόπους όπως είναι η παραμέληση, όπως είναι η άσχημη αντιμετώπιση. Μπορεί να είναι δε πολύ επίπεδη και όσον αφορά την έκφρασή της είτε από μεμονωμένα άτομα είτε και από τις κυβερνήσεις. Το σημαντικό σημαντικό είναι ε, οι Ρωμά να έχουν είσοδη και η ε, πρόσβαση ε, σε όλες τις υπηρεσίες. Να μην τους αρνούμεθα την πρόσβαση αυτή. Να μην δημιουργούνται προγράμματα διακριτικής μεταχείρισης. Να μην χρησιμοποιούνται άσχημα τα, και, τα κονδύλια τα οποία αφορούν τους Ρώμα. αντιαθυγκονισμός μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και στον τρόπο λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ε, θετική επίδραση στη ζωή των Ρωμά, εν τέλει δεν ε, ε, φτάνουν μέχρι αυτού. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι μεγάλες προκλήσεις των Ρωμά, οι οποίοι έχοντα υποστεί επί αιώνε πολλών ειδών καταπίεση και διακριτική μεταχείριση, έχουν πλέον το δικαίωμα να, έχουν, να απολαμβάνουν οι, δύο επίπεδου προστασία με τους ε, άλλους ε, πολίτες. Τους τελευταίους μήνες κάναμε πολλά. Οργανώσαμε ε, εργαστήρια για να δούμε τις διάφορες μορφές αντιαθηγανισμού. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις Ρωμά ή φιλικές προς τις Ρωμά που δουλεύουν δηλαδή υπέρ των Ρωμά. Ήρθαμε σε επαφή επίσης και ανταλλάξαμε απόψεις με διεθνεί οργανισμούς καθώς επίσης και με τους σκιώδει ε, εισηγητέ. Ε, έλαβα υπόψη μου όλα τα στοιχεία τα οποία ε, μου μετέδωσαν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την βοήθεια της γραμματέως της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών χωρίς την βοήθεια της οποίας δεν θα μπορούσα να είχα ολοκληρώσει την εργασία μου. Λάβαμε επίσης υπόψη και τα τελευταία ευρήματα της πρόσφατης μελέτης για το θέμα αυτό. Ε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε τα διάφορα πρόσωπα του ανθιγανισμού από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέχρι την ευρεία και διαδεδομένη ε, διακριτική μεταχείριση από το θέμα της, ε, των απάτριδων μέχρι το θέμα της ένταξης των Ρωμά στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε υποβάλει πολλά ερωτήματα στην Κομισιόν και στο ε, Κοινοβούλιο καθώς επίσης και στις εθνικές κυβερνήσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αμοιβαία, να οικοδομηθεί μάλλον αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των Ρωμά ε, και, γι αυτό, και των υπολείπων. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από την Κομισιόν να δημιουργηθεί Επιτροπή Συμφιλίωσης Ε, και επίσης να υπάρξει μια επίσημη λευκή βίβλος ε, που θα αναφέρεται ακριβώς στο ιστορικό της ε, ε, της δίωξης και της απομόνωσης ε, περιθωριοποίησης των Ρώμα. Ε, παράλληλα ζητώ από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν, να συστήσουν επιτροπές, εθνικές επιτροπές συμφιλίωσης με το ίδιο θέμα. Ως δεύτερο θέμα πρέπει να πω ότι με προβληματίζει ιδιαίτερος ότι σημαντικά προγράμματα όπως ας πούμε αυτά των διαφορετικών ταμείων ταμείων ξεχνούν ε, τους Ρωμά. Γι' αυτό ζητώ από το ελεγκτικό συνέδριο ε, να μελετήσει προγράμματα όπως το Erasmus Plus, εκπαιδευτικά και άλλα, ε, καθώς επίσης και την ακριβή χρήση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση με το ίδιο θέμα. Επίσης, ε, ε, καλεί τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να ε, ληφθούν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση κακής χρήσης των ταμείων. Επίσης, θα θέλουμε να αναγνωριστεί ο ρόλος συγκεκριμένων οργανισμών στην παρακολούθηση του φαινομένου του αντιαφρικανισμού. Ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και αυτό είναι το τρίτο μου θέμα, ε, εκφράζουμε την ανησυχία μας ε, γιατί τις περισσότερες φορές οι Αθήγανοι αποκλείονται από οποιαδήποτε από οποιαδήποτε κρατική διαδικασία. Το πρόβλημα δε είναι ακόμα πιο έντονο στην περίπτωση των απάτριδων. Επίσης καταδικάζουμε τα κράτη-μέλη τα οποία, ε, τα οποία έχουν ε, διακριτικούς τρόπους ε, καταγραφής των Ρωμά. Γι' αυτό, τον, γι αυτό ακριβώς καλό τα κράτη-μέλη να πάρουν αμέσως διαφορετικά μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουν η ισότιμη καταγραφή των Ρωμά στις αρμόδιες αρχές. Ταυτόχρονα δε ζητώ από την Κομισιόν ε, να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη ε, και να ε, παράγει δεσμευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις των χωρών που δεν αναγνωρίζουν ισότιμη πρόσβαση των Ρωμά στη δικαιοσύνη κλπ. Επίσης ζητούμε μέχρι το 2020 να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές πολιτικές, στρατηγικές και μέτρα ε, ενσωμάτωσης των Ρωμά και καταπολέμηση του ανθιγανισμού. Επίσης, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, την παροτρύνω δηλαδή, ε, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους Ρωμά, καθώς επίσης και να καταγράψει όλα τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Επίσης, να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα ε, προβλήματα τα οποία είναι συγγενή με την αθηγανοφοβία. Ε, αυτά είναι τα τέσσερα κύρια στοιχεία τα οποία με απασχόλησαν στην έκθεσή μου η οποία οπωσδήποτε θα συμπληρωθεί και από ε, ε, τροπολογίες. Ε, μια και η κατάσταση των Ρωμά είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, θα ήθελα να λάβω ένα καλό input ε, από τους ε, ε, συναδέλφους και προσδοκώ λοιπόν και από τους σκιώδεις και από τους υπολείπους να, με, να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Μέχρι τώρα στις συναντήσεις με τους σκιώδεις τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά και επομένως προσδοκώ καλά αποτελέσματα από αυτήν την συνεργασία πάνω σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλία θα ήθελα βεβαίω να ευχαριστήσω και την Ρίτα Φόρμπερ με την οποία να δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά καθώ επίση και τον Ινίγκο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζουμε ότι σα απασχολεί πολύ αυτή η έκθεση και είναι μια έκθεση ιδία πρωτοβουλία που αξίζει πραγματικά την προσοχή των συναδέλφων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω του συναδέλφου μου εδώ και ενδιαφέρονται για το θέμα γιατί πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Ήταν ενδιαφέρον ο κατάλογος ε, που αναφέρατε και η έκθεση αυτή νομίζω πρέπει να αναφέρει ποια είναι αυτά τα κενά που υπάρχουν ακόμα στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Να πω λίγο κάτι. Ναι, επειδή ευχαριστήσατε το προσωπικό, ε, επειδή συνήθως όταν τα λέω λείπουν όλοι να τους ευχαριστήσω τώρα το προσωπικό μας ε, με τις Πριν εξαφανιστούν όλοι αύριο, να ευχαριστήσω την γραμματεία, όλη την ομάδα. Πριν ε, πέσετε λοιπόν αύριο και πάτε διακοπές. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο κάνετε. σωράγε Σας ευχαριστώ λοιπόν. Περνάμε τώρα στους πολλούς συναδέλφους που θέλουν να σχολιάσουν το σχέδιο έκθεσή σας. Ε, ξεκινάμε τον κύριο Τράκη που είναι σκιώδης εισηγητής από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ. Κλοντ, ε, σας ευχαριστώ για το ότι ασχοληθήκατε με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι ευρύτατο νομίζω και θα ήθελα να ζητήσω και το σχέδιο αυτό από την κυρία Ευρωβουλευτή. Εγώ θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική η έκθεση, η κυρία Πόστο έχει κάνει διάφορες συστάσεις ε, τις οποίες μπορώ να στηρίξω εξ ονόματος του ΕΛΚ Πούμε λίγο για το ότι δεν έχουμε χρονικό περιθώριο μεγάλο, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. έχω κάποιες παρατηρήσεις που θα υποβάλω τροπολογίες. Θα ήθελα να πω το εξής όμως σύντομα. το έγγραφο αυτό δεν είναι πλήρως ισορροπημένο. Μιλάμε για την ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά πρέπει να υπάρξει και η ανάγκη αυτοοργάνωσης ε, της κοινωνίας ε, των Ρωμά για τις ε, ευθύνες της intelligentsia, θα έλεγα, της κοινότητας των Ρώμα πρέπει να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Η άλλη ανισορροπία είναι ότι το έγγραφο είναι πολύ δυτικό θα έλεγα. Θα αναφέρω τρία κράτη-μέλη ε, χωρίς να τα κατηγορώ απλά να σας δείξω ότι το θέμα αυτό έχει εστιαστεί κυρίως στην ανατολική πλευρά, στην Ρουμανία, Βουλγαρία και στη χώρα μου την Σλοβακία όπου το ποσοστό των Αθήγανων είναι υψηλότερο. Στις τρεις χώρες αυτές έχουμε ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει στη, σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα των καταβλισμών. Είναι, κύριε Πρόεδρε, έσχος ε, το ότι ανεχόμαστε αυτές τις αναξιοπρεπείς συνθήκες για Ευρωπαίους πολίτες ε, τις συνθήκες αυτές διαβίωσης. Ε, δεν το λέω θεωρητικά. Ήμουν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχω εμπειρία από πρώτο χέρι ότι το θέμα δηλαδή των ε, καταβλισμών ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ξεχωριστό και να έχει δική του χρηματοδότηση από τα διαφορετικά ταμεία. Και θα πρέπει ακριβώς ε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Κατόπιν έχουμε το θέμα της ενεργείας. Η ψαλίδα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Η κοινωνία απαιτεί όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Και βλέπουμε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης ε, των Ρωμά υστερεί. Και πάλι αυτό είναι πρόβλημα κυρίως των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποια προγράμματα κατά προτεραιότητα που έχουν δοκιμαστεί αλλά δεν έχουν εισαχθεί σε εθνικό επίπεδο. Συμφωνώ με, τους, με την συνάδελφο την κυρία Πόστ ότι το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης και της εκπαίδευσης των μηνοτήτων είναι κάτι το πολύ ε, σοβαρό. Φοβούμαι ότι η χώρα μου, η Σλοβακία, είναι μια χώρα όπου είχαμε ένα κόμμα που πλέον είναι στον κυβερνητικό συνασπισμό που κατέβηκε με αντιαθηγανική ε, προπαγάνδα. Και βεβαίως ε, ο Πρωθυπουργός της ε, Σλοβακίας έκανε και κάποιες παρατηρήσεις κατά τον Ρωμά για να Αποσπά την προσοχή από ένα σκάνδαλο τότε διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Σόφι Νετφέλντ. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω σύντομη δήλωση εκ μέρους της Σιλία Βίξτρομ, η οποία ε, προεδρεύει στην Επιτροπή Αναφορών αυτή τη στιγμή. Για πάνω από 500 χρόνια οι Ρωμάνοι στην Ευρώπη είναι κομμάτι της Ευρώπης αυτούς τους αιώνες αντιμετώπισαν αποκλεισμούς και διακρίσεις. Σε ένα από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της ευρωπαϊκής ιστορίας, οι τσιγκάνοι βρήκαν το θάνατο στους αλαμούς αερίων. Ακόμη και σήμερα, οι διώξεις τους είναι εκτεταμένες στην Ευρώπη. Θα ήθελα να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους συνεισηγητές, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ορθώσει τη φωνή του υπέρ των τσιγκάνων. Μετά από αιώνες δολοφονιών και καταπίεση ήρθε η ώρα να σκεφτούμε διαφορετικά και η Ευρώπη να κάνει αυτό που πρέπει. Είναι καιρό να αντιμετωπίσουμε την ιστορία μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ενώπιον της ιστορίας. Ευχαριστώ. Α, ε, εκ λοιπόν σκιώδου της Άλντε. Πολύ ωραία. Ε, και τώρα όσον αφορά την γνώμη της Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιόρκ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη κυρία Αλμπή, η οποία είναι σκιώδη, αλλά δεν μπορεί να παρευρεθεί. Μου ζήτησε να σα παρουσιάσω την απόψη τη. Θα μιλήσω αγγλικά εν συνεχεία. Πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ για το εξαιρετικό έργο και τη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και δι' με την κοινωνία των πολιτών και τους ακτιβιστές. Η έκθεση αποτελεί σημαντικό σταθμό στις προσπαθίες μας. Πρέπει να ορίσουμε βεβαίω τον αντιαθήγανισμό όπως το ονομάζουμε. Το κείμενο είναι μια καλή βάση για μελλοντική νομοθεσία κατά των κηρύγματων μίσους που δεν καταγγέλλονται παρκώς όταν γίνονται κατά Ρωμά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ένα χειρό μήνυμα εν ώψη της διαμόρφωσης του νέου πλαισίου για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Οι διακρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διακρίσεις, ως ένα πολιτικό διαρθρωτικό πρόβλημα των κοινωνιών μας εν το σύνολο τους. Λόγω αυτού του δομικού ρατσισμού δεν έχει εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπαρκής Νομοθεσία ούτε αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Σε μερικά κράτη-μέλη τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται για την κατεδάφιση οικισμών ή την κατασκευή σχολείων που ουσιαστικά αποτελούν γκέτο. Πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν για την καταπίεση, την μυσαλλοδοξία και να λάβουμε υπόψη μας την ειδική κατάσταση των Ρωμά ΛΟΑΔ. Πρέπει να προστατεύσουμε επίσης το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση. Πιστεύω επίσης ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της μυσαλλοδοξίας είναι η εμπλοκή των δημοσίων αρχών του κράτους. Ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι σε θέση να προαγάγει την ισότητα. Τα δικαιώματα πρέπει να τη χάνουν εγγύσεων από το κράτος. Όπως γίνεται άλλωστε με την ε, εκπαίδευση, την στέγη κλπ. Χωρίς τον δημόσιο τομέα δεν θα μπορούσαμε ποτέ να εγγυηθούμε τα δικαιώματα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ, ποτέ να τα προστατεύσουμε. Συνεπώς έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι ορισμένα χάσματα, ορισμένες διαφορές ε, διονγκώνονται αντί να συρρυκνώνονται. Θα υποβάλουμε σχετικά κάποιες τροπολογίες, θα συνεργαστούμε όμως βεβαίως ευχαρίστως με την εισηγήτρια και τους κοιόδης και να συνεχίσω στα σφυδικά για τα σχόλια της Επιτροπής Γυναικών. Στην Επιτροπή γυναικών αποφασίσαμε ότι θα υποβάλουμε τροπολογίες για να τονίσουμε την γυναική διάσταση. Υπέρ των Ρωμα γυναικών και κοριτσιών. Αργότερα αύριο θα ψηφίσουμε επιθυμάτων που αφορούν την εκπαίδευση γυναικών και νεαρών κοριτσιών μεταξύ άλλων εδώ βεβαίω μας ενδιαφέρουν οι γυναίκες Ρωμά και το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για το σώμα τους. Το θέμα είναι μεταξύ άλλων και σεξουαλικής υγείας. Εδώ πρέπει να αρθώσουμε τη φωνή μας εν ώψη του τελικού κειμένου. Είναι θέμα το οποίο θα και στην Επιτροπή Ισότητας. Και τώρα... Ευχαριστώ. Ε, θα μιλήσω κι εγώ σου ειδικά, γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το εξαιρετικό αυτό έγγραφο και ξέρω πως υπάρχουν και άλλα πολλά που δεν μπόρεσαν να χωρέσουν στην έκθεση λόγω των κανόνων που έχουμε για το μήκος των εκθέσεων και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε με την Σωραία και θα τα βάλουμε μετά στις τροπολογίες είναι μια εξαιρετική βάση και νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε πολλά από την Σοράγια. Λοιπόν, έχουμε διαφορετικές ομάδες εδώ πέρα, εθνικές μειονότητες θα έλεγα. Μιλάμε για Ρωμά οι οποίοι έχουν δικαιώματα στην χώρα μας από άλλες χώρες και πέρα από τους Σουηδούς Ρωμά έχουμε και Φιλανδούς Ρωμά αλλά και πολλούς από την πρώην Γιουγκοσλαβία που ζουν στην Σουηδία εδώ και καιρό αλλά συχνά αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Επίση έχουμε και άλλους μετανάστες από την Ένωση που έφτασαν τα τελευταία χρόνια, πολλοί που ζητιανεύουν στις πόλεις μας και στην Σουηδία είναι κάτι το καινούριο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους, έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως και όλοι οι υπόλοιποι κοινοτικοί μετανάστες. Έχουμε όμως και αρκετούς ετούντες άσυλο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωμά όμως, που ήρθαν στην Σουηδία πριν από λίγα χρόνια. Π.χ. πριν από λίγα χρόνια ήταν Σέρβοι, Ρωμά, που ζητούσαν άσυλο. Και παρά το ότι ήταν λίγοι, ε, δεν τους ε, επιτράπει να μείνουν και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Επίσης ε, πρέπει να δούμε το πώς έχει η κατάσταση στις υποψήφιες χώρες. Στην Τουρκία π.χ. έχουμε την έκθεση πρόοδου που την είδαμε στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί πέρα υπάρχει ένα εδάφιο που μιλάμε για τους Ρωμά στην Τουρκία. Κάτι λοιπόν πρέπει να πούμε και για το τι γίνεται στις υποψήφιες χώρες. Υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε το τι λείπει από την έκθεση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που λείπουν και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Σοράγια, θα κάνουμε και τις δικές μας προτάσεις πέρα από αυτά τα οποία είπε η Σοράγια και θα εστιάσουμε στους μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ετούντες ασύλου. Σας ευχαριστώ ο κύριος Νίντερ Μιουλαρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Σοράγια. Άρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για την Επιτροπή μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα γιατί γνωρίζουμε ότι η Ρωμά είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα είναι και πολίτες της Ένωσης, όπως είμαστε κι εμείς. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως η κατάσταση στα κράτη-μέλη δεν είναι ίδια. Ε, νομίζω πως η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δείχνει διαφορετικά, διαφορετική κατάσταση και Τσάκη αναφέρθηκε στο ότι σε κάποιες χώρες έχουμε διαφορετική κατάσταση. Πρέπει επίσης να τονίσουμε την κοινωνική ένταξη, τον ρόλο της κοινωνικής ένταξης, την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στέγης κτλ. Πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά άκουσα την Μάλιν γιατί αναφέρθηκε στην κατάσταση των γυναικών Ρωμά, άλλο πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερο και πρέπει και εκεί να επικεντρωθούμε και τέλος κάτι που μπορεί να σκεφτεί ίσως η Σωράγια, έχουμε και καλά παραδείγματα κοινωνικής ένταξης, ε, πρέπει να τα λέμε και αυτά και να συγκρίνουμε καλές πρακτικές και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε το πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών Ρώμα και τις ε, κατευθυντήριες γραμμές καταπολέμησης των διακρίσεων για να έχουμε έτσι ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ σωράγια για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Συγγνώμη, είχα αφήσει το μικρόφωνο ανοιχτό. Λοιπόν, συμφωνώ πλήρως ότι τα θετικά μοντέλα ένταξης είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα ε, συγγνώμη, η Σωράγια δεν πρέπει να σχολιάζω υποτίθεται την έκθεση ως ε, πρόεδρος, αλλά το ξεχνάμε αυτό συχνά στις εκθέσεις μας. Και σταματάω εδώ. Άννα Γκόμες. Στη χώρα μου την Πορτογαλία. Σήμερα. Είχαμε μία ανεπανάληπτη απόφαση που έλαβε ο εισαγγελέας που κατηγόρησε ένα ολόκληρο αστυνομικό τμήμα επειδή επιτέθηκε σε μια ομάδα, σε μια γειτονιά, σε μια ομάδα νεαρών, κυρίως μαύρων. Ταυτόχρονα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την κηδεία ενός Πορτογάλου πολίτη, ενός Αθήγκανου, που δεν επιτράπει να ταφεί στο νεκροταφείο. Λόγω του ρατσισμού του Δημάρχου. Απαράδεκτα πράγματα, ρατσισμός. Μιλάμε για μια χώρα όπου ε, το κράτος ε, με στήριξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων προσπαθεί να εντάξει τους Ρωμά αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το στίγμα αυτό. Οπότε, σωράγια, ελάτε στη χώρα μου για να επισκεφτείτε κάποιες ε, κοινότητες όπου εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα το στίγμα του ρατσισμού, όπως ε, φάνηκε από τα γεγονότα που ανέφερα. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Πορτογαλία. Πραγματικά έχω μείνει άναπτη από αυτό το οποίο είπε ο Σλοβακός συνάδελφος. Επισκέφθηκα τη Σλοβακία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας όταν συζητούσαμε την απαράδεκτη νοοτροπία της χώρας αυτής ε, όσον αφορά την αντίδρασή της στην προσφυγική κρίση. Ε, είδα τα επιχειρήματα που ακούστηκαν στις συζητήσεις μαζί μου. υπήρχε ε, συστηματική πολιτική στιγματισμού των Ρωμά και των ε, προσφύγων. Ε, τους έβλεπαν μόνο ως απειλή τρομοκρατίας. Πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση το ότι είχαμε τέτοια ρατσιστικά επιχειρήματα κατά των ευρωπαϊκών αξιών. Οπότε σύμφωνο πλήρω με τα συμπεράσματα εδώ της ε, εισηγήτριας και αντί για ένα οικονομικό και πολιτικό πρόγραμμα χρειαζόμαστε κάποια συμφιλίωση και συνοχή και να εκπαιδεύσουμε τους νέους έτσι ώστε οι νέοι οι νέοι Ρωμά να μην υφίστανται διακρίσεις όπως σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει τον λόγο. Λοιπόν, να προσθέσω και εγώ κάτι σωρά για μια ερώτηση. Θυμάμαι κάποιες εκθέσεις για τις μειονότητες που είχαν γραφτεί εδώ και χρόνια και βεβαίως υπάρχει εδώ και χρόνια η δουλειά που γίνεται για τα ζητήματα αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Το θέμα του πού συγκεντρώνονται οι κοινότητες των Ρωμά που είναι σε λίγες χώρες αλλά υπάρχουν κοινότητες ε, Ρωμά και σε δυτικές χώρες που είναι πιο διασπαρμένες. Κατά την άποψή σου ε, θα πρέπει να δούμε τις ανάγκες αυτών των πιο διασπαρμένων κοινοτήτων που ίσως υφίστανται διαφορετική διακριτική μεταχείριση. Ε, ε, θα κοιτάξει τα πιο στρατηγικά ζητήματα στις τρει τέσσερι χώρες όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόθεσή σου, γιατί κατά κάποιον τρόπο ε, δεν θέλω να υπάρχει αυτό το διέρη και βασίλευε και να λέμε ότι έχουμε μία έκθεση δυτική που κατηγορεί την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Γιατί όταν έγραψα εγώ έκθεση για τις μειονότητες αυτή ήταν η κατηγορία Οπότε αναρωτιέμαι έτσι πώς ε, έχεις χαράξει την στρατηγική της έκθεσης σου. Γιατί υπάρχει πράγματι μεγαλύτερη συγκέντρωση της κοινότητας σε κάποιες ε, χώρες. Και, αλλά κάποια από αυτά τα ζητήματα, όπως είπαμε, ε, ισχύουν και για την ε, Δυτική Ευρώπη, όπως ακούσαμε, λόγω της κρίσης των προσφύγων και άλλων θεμάτων. Αν θέλεις, μπορείς να απαντήσεις στα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Κλοντ, θα μιλήσω και εγώ σου ειδικά. Λοιπόν, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τα σχόλια που έκαναν. Στην Μάλιν να πω ότι με ιδιαίτερος ευγνώμων για την προσθήκη που πρότεινες για την κατάσταση γυναικών ε, και κοριτσιών. Ε, το είχα σκεφτεί. Ε, δεδομένου όμως το ότι έχουμε περιορισμού στο κείμενο, ήξερα πως κάποιοι από την Επιτροπή ΦΑΜ θα το πρότειναν. Ξέρω πως έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και σκεφτόμαστε τα ίδια βεβαίως, το μιλάμε για τα δικαιώματα όλων. Προφανώς ε, είναι ιδιαίτερος ευπαθής οι γυναίκες ε, Ρώμα. Στον ε, να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει στην έκθεση μια αναφορά για τους Ευρωπαίους πολίτες Ρωμά που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις χώρες τους ε, και να πάνε αλλού και βρίσκονται στους δρόμους να ζητιανεύουν. Ε, πάνε δηλαδή για να βρουν δουλειά, αλλά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και όσοι φεύγουν από τις χώρες τους ε, δεν έχουν βεβαίω ούτε τις εμπειρίες, ούτε την εκπαίδευση και δυστυχώς συχνά καταλήγουν ε, να ζητιανεύουν έξω από τα καταστήματα, στους δρόμους στη Σουηδία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, πρέπει να καλυφθεί αυτό στην έκθεση. Και βεβαίως ε, όταν προσπαθούμε να έχουμε κάποιους κανόνες για την ελευθερία μετακίνηση, δεν σκεφτόμαστε τους Ρωμάνους, είχαμε σκεφτεί ίσως ε, θα είχαμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ακριβώς ίδιες οι συνθήκες για όλους. Πολλοί δεν έχουν την κάρτα ασφάλισης υγείας. Υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που θα ήθελα να δω όταν μιλάμε για τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας, όπου δεν ε, έχουμε σκεφτεί ε, το ότι υπάρχει μια ομάδα τόσο πολύ εκτός των δομών της κοινωνίας που δεν τους ε, σκεφτόμαστε ή όταν μιλάμε για την ελευθερία μετακίνησης είτε για τις οδηγίες κατά των διακρίσεων κτλ. Αυτό προσπαθώ να αναδείξω. Αυτή η ιστορία του αντιαθηγανισμού που πρέπει να το δούμε εάν είναι να έχουμε κάποια πραγματική ένταξη στην κοινωνία. Πρέπει, πώς να το πω, Πρέπει να σταματήσουμε να ε, σκεφτόμαστε και να δίνουμε ασπιρίνες ε, για το θέμα. Έχαμε και το ψήφισμα για τον αντιαθηγανισμό. Έχουμε κάνει την διάγνωση. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα δράσουμε. Ε, πρέπει να υπάρχει μια λειτουργική προσέγγιση Χρειαζόμαστε λοιπόν μια επιτροπή αλήθειας, μια διαδικασία συμφιλίωσης, όπως είπε η Τζάκη. Ε, πρέπει η Ρώμα να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Πράγματι, αλλά όταν κάποιο είναι τόσο πολύ εκτός ε, των ε, δομών και μιλάω και από την εμπειρία μου, εάν η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου είναι ότι είσαι άλλη κατηγορία πολιτών, ότι δεν αξίζει τίποτα γιατί αυτό σου λέει κοινωνία επί αιώνε, τελικά έχει εγγραφεί στην ίδια σου την ταυτότητα και την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Πρέπει λοιπόν να το φροντίσουμε αυτό. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι, να υπάρξει εμπιστοσύνη και να ε, προχωρήσουμε παραπέρα. Εγώ η ίδια μέχρι πριν από 15 χρόνια θεωρούσα εαυτήν ε, ως ε, πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Και δεν μπορούσα να δεχτώ το πώς ήταν διαμορφωμένη η κοινωνία, γιατί θεωρούσα ότι δεν είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας και χρειαζόταν χρόνια για να το ξεπεράσω. Ζούσα σε μια κοινωνία άδικη και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ήθελα να συνεισφέρω, είχα αυτά τα ενδιαφέροντα, μπορούσα να συνεισφέρω στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας και έφτασε κάποια στιγμή η μέρα που συνειδητοποίησα και ε, το δούλεψα πάρα πολύ μέσα μου αυτό που είπα ότι όχι, είμαι μια, μια πολίτης πρώτης κατηγορίας. Δεν είμαι ε, ε, χειρότερη ή καλύτερη από τους άλλους και θα συνεισφέρω. Αυτή ήταν μια αίσθηση. Ε, αφού είχα γεννήσει τέσσερα παιδιά, ε, θα έλεγα μετά από τα παιδιά μου ήταν το εντονότερο συνέστημα που είχα νιώσει. Και νομίζω οι περισσότεροι Ρωμά έτσι αισθάνονται. Οι περισσότεροι γονείς Ρωμά θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα <coughs> θετική για τα παιδιά τους. Θένε να έχουν μια θετική συνεισφορά να λένε στα παιδιά διαβάστε, διαβάστε, να πάρετε καλούς βαθμούς, να πάρετε καλούς βαθμούς, να περάσετε στο πανεπιστήμιο, να πάτε καλύτερα στη ζωή σας. Αυτό που θέλουν όλοι οι γονείς ε, για τα παιδιά τους. Και ε, θα έλεγα ακόμα και αυτοί που είναι στο δρόμο και ζητιανεύουν. Είναι στο δρόμο και ζητιανεύουν για να μην έχουν τα παιδιά τους τη ζωή που είχαν αυτοί. Τα λεφτά πηγαίνουν κατευθείαν ε, σε φαΐ και ένδυση για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Η στρατηγική λοιπόν είναι να υπάρξει ενημέρωση σε όλα τα κράτη-μέλη για τον αντιαθηγανισμό τους. Και βέβαια αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά το κοινό σημείο είναι ο αντιαθηγανισμός που οφείλεται στην πολιτική, οφείλεται στις δομές, οφείλεται στην ανάληψη ευθύνης ε, και στο ότι οι χώρες θα πρέπει να βλέπουν τους πολίτες, τους Ρωμάς τους πολίτες και να το αντιληφθούν αυτό και οι δημόσιες διοικήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια αυθαίρετη κατανομή. Και σε μια δημοκρατική κοινωνία αυτό έχουμε. Ε, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, επιρροή από την κορφή της κοινωνίας σε όλα τα στρώματα και ελπίζω η έκθεση αυτή να καλύψει τις συναισθηματικές αλλά και τις διανοητικές ε, πτυχές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές και νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και να προσπαθήσω να περιλάβω όλες τις απόψεις από μικιό από τους σκιώδεις και σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ Σουράγια και τους και Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 18 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την συζήτηση αυτή και τώρα περνάμε στην κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ένωση. Πριν από ένα έτος η Κομισιόν παρουσίασε το δεύτερο νομοθετικό πακέτο για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που είχαμε και έναν κανονισμό σχετικό Ξέρετε συνάδελφοι ότι πρόκειται για ένα φάκελο νομοθετικής προτεραιότητας ε, υπήρχε το πολίτικο σήμερα είχε έναν τίτλο που έλεγε «Μετανάστευση 1596 τροπολογίες». Αυτό είναι ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα ακολουθήσουν και άλλες. Ε, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την εισηγήτρια Λόρα Φεράρα που παρουσίασε στις 29 Μαΐου το σχέδιο έκθεση. Σήμερα θα γίνει μια πρώτη συζήτηση του αριθμού αυτού των τροπολογιών. Λοιπόν, επειδή καθυστερούμε, θα δώσω τον λόγο στην Λόρα αμέσως για να έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο. Έχετε τον λόγο. Λάουρα Φεράρα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων ομάδων και τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει. 1600 ε, ε, ε, υποβληθεί στις τροπολογίες και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει σαφώς και την πολιτική ευαισθησία αλλά και την περιπλοκότητα του θέματος που αφορά αυτή την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κοινή διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο κάναμε μια πρώτη επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να δούμε πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τι υποβληθήσει τροπολογίε και να δούμε ποιε θα μπορούσαν να είναι οι πολιτικές πρωτο... προτεραιότητες των διαφόρων ομάδων. Συζητήσαμε επίση και τη μεθοδολογία της εργασίας ε, που ε, θα ακολουθήσει. Ε, σε μια πρώτη εξέταση των τροπολογιών μου προκύπτουν ορισμένα κεντρικά στοιχεία τα οποία όμως ε, οι διάφορες πολιτικές ομάδες αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο και επομένως ε, εγώ θα εργαστώ με τρόπο ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός συμβαστικών τροπολογιών έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να υποστηριχθεί από όσο γίνεται περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ήδη ε, φαντάζομαι ότι ε, οι τριμερείς διάλογοι και οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο θα είναι μάλλον περίπλοκες και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει σταθερή και ευρεία συνενέσεως θέση. Πρόθεσή μου ε, και ελπίδα μου είναι βεβαίως ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε μέχρι το τέλος ε, τρέχοντος έτους τη θέση του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν ε, και οι συζητήσεις μετά από την αρχή του επόμενου χρόνου. Το Συμβούλιο όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα διαμορφώσει θέση. Οι εργασίες εξ όσων επιβεβαίωσε και η αρμόδια επίτροπος της Προεδρίας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών προχωρούν με πολύ βραδύ ρυθμό. Υπάρχουν βεβαίω σημαντικέ ε, διαστάσει ε, όσον αφορά τι διάφορε πολιτικέ ε, ομάδε. Αναφέρομαι στο κατά πόσο θα πρέπει η διαδικασία αποδοχή να είναι υποχρεωτική ή όχι. Επίση το βάρο το οποίο θα πρέπει να δώσουμε στι ασφαλεί χώρε ή τι ασφαλεί χώρε προέλευση. Θα πρέπει σε όλε αυτέ τι περιπτώσει να καθορίσουμε εάν θα διατηρήσουμε τον υποχρεωτικό υποχρεωτικό χαρακτήρα ή εάν αντιθέτως θα δώσουμε την δυνατότητα στα κράτη-μέλη ε, να εφαρμόσουν ή όχι ε, τις ε, περιπτώσεις αυτές. Επίσης υπάρχουν και άλλα σημεία επί των οποίων θα πρέπει να βρούμε αποδεκτή από όλους συμβιβαστική λύση. Ωστόσο, ο κεντρικός στόχος είναι ε, η ε, πρόσβαση στην προστασία, στη διεθνή προστασία να παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ετούντες άσυλο, ενώ ταυτόχρονα ε, θα να προβλέψουμε μια διαδικασία όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και χρονικά αλλά και από άποψη κόστους. Δεν θα ήθελα να υπάρξουν νέες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις οι οποίες θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές υπάρχουν σημεία επί των οποία ε, είναι πιο κοινέ ε, οι θέσει ε, των πολιτικών ομάδων. Επ' αυτών λοιπόν των σημείων ευελπιστώ ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα και θα επιτύχουμε κοινέ θέσει. Αναφέρομαι στην βελτιστοποίηση των προθεσμιών στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας, την κοινή αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου. Εδώ έχουμε ρεαλιστικές πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη και είναι γεγονός ότι θέλουμε να ε, μικρύνουμε τους χρόνους, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει ο σεβασμός ε, των πραγματικών καταστάσεων ε, που αντιμετωπίζουν οι μεμονωμένε χώρε μέλη να είναι συγκεκριμένοι. Οι διαδικαστικές υποχρεώσεις των ετούντων άσυλο οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύπτονται με ταχύτερες διαδικασίες. Εγώ ως εισηγήτρια σχετικά με αυτή την πρόταση κανονισμού μέσω της υποβολής κάποιων τροπολογιών θέλησα να διευκρινίσω κάποια στοιχεία του σχεδίου εκθέσεώς μου, τα οποία μου είναι ιδιαίτερος προσφυλή ε, ιδίω τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να καθορίσουν ε, ε, ασφαλή τρίτη χώρα. Επίσης, την δυνατότητα και τις διαδικασίες έτσι ώστε να αφαιρεθεί μια χώρα από τον κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης. Επίσης έχω προβλέψει σε όλες τις περιπτώσεις ε, προσφυγής ε, αυτόματη ανακλητική διαδικασία της ε, έφεσης έτσι ώστε επίσης να σταματήσουν οι διαρκείς παραβάσεις. Εγώ θέλησα να άρω την αυτόματη ανακλητική ανακλητική, α, τη αυτόματη ανάκληση της διαδικασίας προσφυγής. Ε, επ' αυτών των σημείων βεβαίως θα πρέπει να προκύψει συμφωνία των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδες εισηγητές ε, για την εργασία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είμαι βεβαία ότι θα συνεχίσουμε ε, σε συνεργατικό πνεύμα, καλό πνεύμα συνεργασία να συζητούμε έτσι ώστε να προκύψει η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέση την οποία εγώ θα κληθώ να υπερασπιστώ στι διαπραγματεύσει με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με του σκιώδει από το ΕΛΚ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πρόεδρε. είμαι σύντομο, λέει ο κύριο Λένερ. γιατί δεν είχα χρόνο να μελετήσω τι 1600 ε, τόσε τροπολογίε. Ναι, τρομερό. Άλλαξα πάντα στο ειστήριό μου. Ε, έχω και βαλίτσα, θα τη γεμίσω με τροπολογίε. θα τι πάρω μαζί μου στι διακοπέ, να τι διαβάσω. Ευχαριστώ, Λόρα, την εισηγήτρια, για τη δουλειά της και για όλες τις ε, συσκέψεις που είχαμε. Ήταν ότι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε για να διαμορφώσουμε μια σαφή θέση εκ μέρους του Κοινοβουλίου, παρά τις ε, διαφορές απόψεων. Θεωρώ ότι η τελική στάση είναι ακριβοδίκη. Το ΕΛΚ και οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει για τις προτεραιότητες. Διαφωνούμε ποια θα είναι η σειρά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει συμφωνούμε επί των προτεραιοτήτων. Ο βασικός στόχος για την διαδικασία ασύλου είναι να είναι μια γρήγορη, απλή διαδικασία, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, έχουμε μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων. Είδα τροπολογίες και από το κόμμα μου, που πραγματικά με κάνω πιστεύω καμιά φορά ότι θα έπρεπε ο κανονισμό να γίνει οδηγία, αλλά σε ορισμένε περιπτώσει εξασφαλίζουμε ευτυχώ αρκετή ευελιξία στα κρατημέλη και στο πλαίσιο του κανονισμού και είμαστε μάλλον εντάξει. Να είμαστε όμω προσεκτικοί. Εάν πάρουμε την απόφαση, αν κρίνουμε ότι τελικώ ο κανονισμό είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη διαδικασία σύλλου κλπ. Να μην δώσουμε υπερβολικά μεγάλο ευρώ ευελιξία στα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένου τομεί, όπω θέλουν μερικέ τροπολογίε, διότι θα οδηγηθούμε σε μια εκ των πραγμάτων σε μια de facto οδηγία. Θα πρόκειται για οδηγία μάλλον παρά για κανονισμό. Και δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αυτό. Είμαι υπέρ λοιπόν του να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίε να είναι παρόμοιε σε όλε τι χώρε, να είναι ίδιε σε όλε τι χώρε, να είναι προβλέψιμε, απλέ, γρήγορε διαδικασίε. Και εν τέλει το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αφενός της προστασίας του δικαιώματος αυτών των ανθρώπων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αιτηθούν άσυλο γιατί φεύγουν από τη χώρα τους λόγω διώξεων, λόγω πολέμου και αφετέρου της ανάγκης αυστηρότητας δηλαδή να μην υπάρχουν περιθώρια κατάχρησης ή απλούστερα, ή απλούστερα κακής χρήσης και αυτό, και σε αυτό αποσκοπούν ορισμένε τροπολογίε. Κάποιοι συνάδελφοι ρίχνουν το βάρο του υπερβολικά ίσω στην ανάγκη προστασία των προσφύγων, αλλά δεν λαμβάνουν επαρκώ υπόψη του αυτού που προσπαθούν να αξιοποιήσουν το σύστημα προ δικό του όφελο. Συμβαίνει αυτό και με τη δική μου ομάδα. Λοιπόν, όταν λέμε για παραδεκτό, όταν λέμε για επιταχυμένη διαδικασία, όταν λέμε για ε, ασφαλής τρίτες χώρες. Ή όταν λέμε για την ειδική κατάσταση των προσφύγων πριν την απομακρυνσή του, στην περίπτωση απόρριψη κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, διαμορφώντα την τελική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλο, να φροντίσουμε οι διαδικασίε να είναι αποτελεσματικέ αλλά και αποδοτικέ. Δεν μου αρέσει η γραφειοκρατία που βλέπω στην πρόταση τη Κομισιόν κατάθεση αίτηση, εξέταση κλπ. Όλα αυτά πηγαίνουν πολύ αργά έτσι πως έχουν τα πράγματα. Το Κοινοβουλίο λοιπόν να γνωρίζει πώς έχει κατάσταση, να γνωρίζει ότι στα σημεία εισόδου οι διαδικασίες δεν είναι εύκολες. Να φροντίσουμε λοιπόν ότι παίρνοντας στα χέρια τον κανονισμό οι άνθρωποι μας επί τόπου θα κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο γρήγορα και ποδορικά μπορούν. Αυτά μόνο ήθελα να αναφέρω. Από εκεί και πέρα προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πίτερ Μίλλερ από τους Σοσιαλιστές. Πρώτον ευχαριστώ την κυρία Φεραρά. Ε, έκανε τεράστιο έργο, πάρα πολλή δουλειά. Εγώ δεν άλλαξα όμω το ειστήριό μου, αγαπητέ συνάδελφε. Έχουμε κι εμείς καταθέσει ένα σωρό τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν τι δικές μας ε, προτεραιότητες, κυρίως όσον αφορά τον συγκερασμό μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ετούντων, έτσι ώστε τα δικαιώματα να την χάνουν βαργούς προστασίας. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματο συνέντευξη σε κάθε περίπτωση για να διαπιστωθεί κατά πόσον το συγκεκριμένο άτομο χρήζει διεθνού προστασία από την καταγραφή του και μετά. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά, ενδεχομένω να υποβάλουν τη σωστή αίτηση. Επίσης να προσέξουμε το θέμα των ασυνοδευτών ανηλίκων, ιδιαίτερα όταν ε, οι κυδεμόνες τους είναι κρατούμενοι. Επίσης, να απαλύνουμε λίγο τις κυρώσεις στην περίπτωση απόπειρας δευτερογενούς μετακίνησης και να διασφαλίσουμε ότι ο ετών έχει αρκετό χρόνο για να προσκομίσει ό,τι λείπει. και η συνέντευξη περί παραδεκτού ε, να είναι προαιρετική και σε καμία περίπτωση να μην προκαθορίζει το αποτέλεσμα της εξαίρεσης της αίτησης. Επίσης ότι περιλαμβάνεται στην έκθεση περί ασφαλαντήτων χωρών να υλοποιείται στην πραγματικότητα και στην πράξη Είμαι επίση βεβαίω ότι η έκθεση αυτή είναι μία από τι πιο σημαντικέ στο πλαίσιο τη ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκή Πολιτική ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου. Εμείς οι σοσιαλιστέ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την κυρία Φεράρα και να τη βοηθήσουμε να στείλει ένα χειρό μήνυμα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πίτερ από την ομάδα ECR. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Φεράρα η ουσία της πρότασης μας βρίσκει σύμφωνος να διευκολύνουμε την διαδικασία και να αποθαρρύνουμε την αναζήτηση ευνοϊκής υποδοχής στην κατάλληλη χώρα, το asylum shopping. Δεν θέλουμε όμως να αποδυναμωθεί ο ρόλος των κρατών μελών στην διαδικασία του ασύλου. Οι τροπολογίες που καταθέσαμε αποσκοπούν στο να δώσουν στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να χειριστούν το θέμα αποτελεσματικά και αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα στα εξή. Το βάρος δεν πρέπει να πέφτει τόσο πολύ στην αλληλεγγύη όσο στην δυνατότητά μας να υποδεχθούμε πρόσφυγες. Οι αρμόδιες αρχές για την εξέταση μιας αίτησης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν έρευνες σε προσωπικά αντικείμενα καθώς και στο περιεχόμενο, το ηλεκτρονικό περιεχόμενο συσκευών. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι ντούντε θα μπορούν να παραμένουν στην επικράτεια του κράτου μέλου. Κάποια κριτήρια πρέπει επίση να βγουν από του λόγου για του οποίου χορηγούμε προστασία. Οι ετούντε επίση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν δωρεάν νομική υποστήριξη στο συγκεκριμένο στάδιο μόνο και όχι σε όλα τα στάδια Επίση, τα κρατημέλη πρέπει να έχουν περισσότερη ελευθερία για να κρίνουν να χρειάζονται πλέον υπηρεσίε, όπω ιατρικέ και ψυχολογικέ υπηρεσίε, υπηρεσίε ψυχολογική υποστήριξη. Επίση στην περίπτωση απειλή κατά τη εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, να υπάρχουν επίση δυνατότητε αντίδραση, να γίνονται ιατρικέ εξετάσεις επίση, και μάλιστα να είναι υποχρεωτικέ για την διευκρίνηση τη ηλικία του ετούντο. Πιστεύουμε επίσης ότι οι προθεσμίες που αφορούν την υποβολή αίτησης πρέπει να γίνουν ακόμη πιο σφιχτές, να προχωράμε πιο γρήγορα. Αυτά προς το παρόν προσβλέπουμε κι εμείς σε περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία με την εισηγητρία και τους συνεισηγητές, τους και οδησηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Σοφία νομίζω εκ αν δεν κάνω λάθος, εκ μέρου ε, Σεσίλια Βίξτρομ, έτσι δεν είναι. Ναι, μου ζήτησε να διατυπώσω κάποιε παρατηρήσεις, αλλά να διατυπώσω πρώτα δύο δικέ μου παρατηρήσεις ως ε, εισηγήτρια την ε, οδηγία για την υποδοχή. Κύριο Λένας μίλησε για την ανάγκη εναρμόνισης. Να μην, και να μην ξαναγίνει ο κανονισμός ουσιαστικά οδηγία να μην υπάρχει υπερβολική ευελιξία. Σύμφωνα οι κανόνε πρέπει να είναι οι ίδιοι παντού. Δεύτερη παρατήρηση, ω εισηγήτρια άλλου κειμένου, θα ήθελα να έχω μια γενική εικόνα των θέσεων που υπερψηφίσαμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Γιατί είπαμε ότι θα ευθυγραμμίσουμε τη θέση μας και τη στάση μας επί διαφορετικών θεμάτων. Αλλά στην οδηγία για την υποδοχή υπάρχει αναφορά στην Eurodac που περιλαμβάνει διατάξεις έως και αντιφατικές αλληλοσυγκρόμενες. Λοιπόν, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ζήτησα από τη γραμματεία να μου δώσει μια γενική εικόνα, μια επισκόπηση των θέσεων που ήδη έχουμε υπερψηφίσει για να έχουμε και ένα μπούσουλα. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε και για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, η θέση της Σεσίλια Βίξτρομ ευχαριστεί την ισχυτρία για την επικοδομητική στάση. Υπάρχει ένα τεράστιο αριθμό τροπολογιών. Πρέπει να δούμε να τις επαναδιαμορφώσουμε σε συμβαστικές. Η Κομισιόν θα βοηθήσει προκειμένου, φαντάζομαι, η διαδικασία να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποδοτική, με σεβασμό πάντα στα δικαιώματα των ετούντων. Δεν συμφωνώ με αυτού που, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, υπέρ του να προστατεύονται μόνο τα ελάχιστα δικαιώματα, τα βασικά δικαιώματα. Η Σεσίλη επίση λέει ότι πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε νομική υποστήριξη, παρουσία δικηγόρου κλπ. Αυτό μα βοηθάει να αποφεύγουμε και λάθη τα οποία έχουν μεγάλο κόστο για του ετούντε. Το σύστημα λοιπόν πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, α πούμε, πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια. Εδώ έχει κατά τη περιοριστεί το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά οι ενδιαφερομένοι έχουν το δικαίωμα άσκησης έφεσης. Η Σεσίλια νομίζω δεν θα εκπλαγεί αν μάθει ότι η καθυστέρηση όλες αυτές τις διαδικασίες θα έχει κόστος το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από το ε, εάν δίναμε δωρεάν νομική βοήθεια από την αρχή. Ε, αυτά τα λέω επειδή ξέρω και το θέμα τη νομική βοήθεια στο πλαίσιο τη οδηγία για την υποδοχή. Η Σεσίλια Βίξτρομ επίση πιστεύει ότι έχει μεγάλη σημασία να συγκεράσουμε ικανοποιητικά τι υποχρεώσει με τα δικαιώματα των ετούντων. Μπορούμε πιο συγκεκριμένα να ζητάμε από του ετούντε να παραμένουν στην επικράτεια του κράτου μέλου, το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να απορρίπτουμε τι αιτήσει του μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να ε, καταχωρήσουν μια διεύθυνση στη συγκεκριμένη χώρα. Να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, λέει και η Σεσίλια, να θεωρήσουμε μια πρακτική στάση με σκοπό τελικά να πάρουμε στα χέρια μας ένα σύστημα λειτουργικό. Ευχαριστώ Σκά Κέλλερ για τους πράσινους. Νομίζω ο συνάδελφος ήταν πρώτα, αλλά δεν πειράζει. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα και βεβαίως ε, και στην προηγούμενη ε, συνεδρίαση εμείς αναφέραμε τις προτεραιότητές μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τέλος, το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή, να είναι τέτοιο που να διασφαλίζει ε, ότι ε, θα έχουν πραγματικά δικαιώματα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αιτούντε άσυλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε βεβαίω υπόψη μα ε, την ε, κατάσταση επιτόπου. Ξέρω ότι πολλοί συναδελφοί αναφέρθηκαν σε καταστάσει όπου κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν στα λόγια, στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, αβάσιμο, α πούμε, αίτηση γιατί έχει έχει προκύψει μια εσφαλμένη διεύθυνση και διάφορα άλλα σχετικά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργήσει καλά το θέμα, αλλά οπωσδήποτε πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι εδώ συζητάμε για ανθρώπους για τους οποίους μια απόφαση ιδίω δε αρνητική απόφαση μπορεί να, έχει, να, να αποτελεί απειλή για τη ζωή τους. Αυτό να μην το λησμονούμε. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην υποβάλλουμε ιδιαίτερα επιπλέον φόρτο στις χώρες για μια de facto ας πούμε να φορτώσουμε στις πλάτες ε, των κρατών αλλά και των ετούντων άσυλο ε, μια δεύτερη διαδικασία υποβολής αιτήματος ε, ασύλου νομίζω ότι και πέρσι και πρόπερσι πολλές χώρες αναγκάστηκαν, ήδη είχαν προβλήματα με την απλουστευμένη διαδικασία, να μην τους επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Ε, τα δικαιώματα των ε, ετούντων ε, άσυλο είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις οποιονδήποτε αλλαγών ή περιορισμών μπορεί να είναι συγκλονιστικές για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θέλουμε να μειωθούν τα δικαιώματά τους, κυρίως στη μετακίνησή τους από τη μία χώρα στην άλλη. γιατί ε, πραγματικά ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι η αναζήτηση ε, δικαιοσύνης και ασύλου. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να θεωρηθεί ότι οι επιταχυμένες διαδικασίες ε, είναι σωστές για ανθρώπους που έχουν προφανώς αβάσιμες αιτήσει, γιατί νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν ε, γιατί για να βρεθεί η μη βάσιμη ε, αίτηση ε, εντός ενός μιας ομάδας είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ας πούμε σε περιπτώσεις σύρων προσφύγων, ναι, εκεί μπορεί οι διαδικασίες να είναι πιο γρήγορες και επιταχυμένες, αλλά όχι σε όλες τις ομάδες. Επίσης υπάρχουν και στοιχεία τα οποία ανέφερα στην συνάντηση των σκιωδών και τα ανέφερα στην εισηγήτρια με την οποία βεβαίως θέλω να συνεργαστούμε καλά και μέχρι τέλους. Ε, είναι όντως δύσκολο να ε, βρούμε το δρόμο μας ανάμεσα σε, διάφορες, ε, σε διάφορους κανονισμούς, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη και όσα αναφέρονται και σε άλλα κείμενα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σκά. Λάουρα. Πριν σου δώσω το λόγο, θα ήθελα να ε, έχω την άποψη της Κομισιόν και της Προεδρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε και την εισηγήτρια αλλά και τις πολιτικές ομάδες που εκφράστηκαν ε, για τις προτάσεις τους. Ε, η ΛΥΜΠΕ βεβαίως έχει προτείνει μεγάλο ρυθμό τροπολογιών που θα μελετηθούν προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένες αντιδράσεις γιατί η αντίδρασή μας σήμερα μπορεί να είναι μονάχα γενική είναι περίπλοκο το ε, ίδιο το εργαλείο ε, και ε, βεβαίω περίπλοκες και οι προσεγγίσεις της εισηγητρίας και των σκιωδών εισηγητών. Είναι βέβαιο ότι η εισηγήτρια θα πρέπει να δουλέψει σκληρά τον επόμενο, το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επιτευχθούν δύσκολες συγκλήσεις μεταξύ σαφώς δισταμένων απόψεων. Πολύ σύντομα να υπενθυμίσουμε τον, ε, την ουσία και τον στόχο της ε, πρότασης της Κομισιόν. Ε, Επελέγει το εργαλείο του κανονισμού κυρίως διότι υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί ένα, ένας χώρος προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ικανός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ετούντων άσυλου έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας να την δεχτούν με τρόπο όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό. Ε, και επίσης με στόχο να διατηρηθούν ε, οι πόροι των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρειάζεται κατά την άποψή μας ένα διαδικαστικό εργαλείο το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ανάγκες των ετούντων διεθνούς προστασίας. Γνωρίζουμε ότι τα εθνικά συστήματα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικύλουν και θέλουμε να αποφύγουμε δευτερογενείς ε, ε, μετακινήσεις μεταξύ αποκλει... Ε, ε, αποκλεινών των εθνικών ε, συστημάτων. Δεν θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα οι αιτούντες άσυλο να επιλέξουν τη μία χώρα αντί, την, αντί γιατί στη μία χώρα μπορεί να υπάρχουν διαδικαστικά πλεονεκτήματα. Θέλουμε εναρμόνιση, θέλουμε επίσης εναρμόνιση των διαδικασιών, θέλουμε και εναρμόνιση των χρονικών προθεσμιών, διευκρίνηση της, του αντικτύπου που μπορεί μπορεί ε, να έχει η χρήση των ε, καταλόγων Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλών χωρών, τρίτων ασφαλών χωρών και ασφαλών χωρών προέλευσης. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και δικαιότερα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και η ε, κατανομή του βάρους μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι δικαιότερη. Πιστεύουμε επίσης ε, ότι με τον τρόπο αυτό ακολουθούμε και το πνεύμα της περσινής δήλωσης ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει περαιτέρω να διευκρινιστούν οι διατάξεις στην οδηγία για την ασφαλή χώρα προέλευσης και για την πρώτη χώρα εισόδου ε, και όλα αυτά διατηρώντας ε, τα απαραίτητα εχέγγυα ε, τα οποία πρέπει να υπάρξουν, δηλαδή ότι κανένας να μην, να μην ξεγλιστράει που να μην έχει πραγματική ανάγκη διεθνούς προστασίας. Νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται και στην πρόταση της Κομισιόν όπου προτείνεται νομική αρρωγή, δωρεάν νομική αρρωγή για όλους τους ετούντες με πολύ μικρό αριθμό εξαιρέσεων. Αυτό από μόνο του όχι μόνο δίνει δυνατότητα στα συστήματά μας να ε, σεβαστούν τα δικαιώματα των ετούντων, αλλά βελτιώνει και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Όσον αφορά συγκεκριμένε τροπολογίες, ε, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να μπούμε σε αυτή τη φάση σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, υπάρχουν πολλές ε, τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική έκθεση. Πολλές τροπολογίες είναι αποδεκτές, αυτές οι οποίες θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, αυτές οι οποίες καλούν σε προσεκτική μεταχείριση και αντιμετώπιση Κυρίω κυρίως ε, όσον αφορά τις ε, διαδικασίες ε, αβασιμότητας της αίτηση, καθώς επίσης και την έννοια της επιταχυμένης διαδικασίας. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λόγια από την Προεδρία. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τον λόγο και την δυνατότητα να σας πούμε πώς έχει το θέμα αυτό και ποια είναι τα επόμενα βήματα στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ επίσης το Κοινοβούλιο, την συγγήτρια και τους κοιότητες εισηγητές για τη δουλειά που έχουν ήδη κάνει. Υπό λοιπόν, την Μαλτέζικη Προεδρία, η εξέταση της πρότασης ε, συνεχίζεται στην ομάδα εργασίας ασύλου και έχουμε σχέδια συμβαστικών προτάσεων που συζητήθηκαν για τα άρθρα στο πλαίσιο της θεματικής προσέγγισης που ακολουθεί η Προεδρία μας. Οι διατάξεις που αφορούν ετούντες με ειδικέ ανάγκες αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δύσκολες ε, όσον αφορά το περιεχόμενο, τον συντονισμό και την συνοχή με παρόμοιες διατάξεις σε άλλες προτάσεις του πακέτου. Ε, αυτήν την έννοια έγινε μια προσπάθεια για να υπάρξει μια ευθυγραμμιστή των διαδικασιών, του χρονοδιαγράμματος, των ρόλων και των διαφορών καθηκόντων. Βασιζόμενοι σε αυτό υπάρχουν ακόμα πολλά άρθρα της πρότασης που δεν έχουν συζητηθεί στην ομάδα εργασίας ασύλου και ιστονική Προεδρία θα συνεχιστούν οι συζητήσεις τη συζήτηση της Εσθονικής Προεδρία θα γίνει ήδη την επόμενη εβδομάδα στην ομάδα εργασίας ασύλου, όπου συζητάμε με... ξεκινάμε τα άρθρα που δεν έχουν συζητηθεί καθόλου και σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση του φακέλου το συντομότερο δυνατόν για να περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση και τελικά να καταλήξουμε σε μια θέση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χρήσιμο αυτό και να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπαν και οι συνάδελφοι να ευχαριστήσουν την Λαούρα Φεράρα, Λάουρα Φεράρα. Λάουρα, αν θέλετε να ολοκληρώσετε, αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, λέει η κυρία Φεράρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου όλους τους και την Κομισιόν και το Συμβούλιο που πήραν το λόγο. Ε, θα ήθελα ε, να πω επίσης ε, ότι εγώ θα προσπαθήσω να διασφαλίσω την μέγιστη δυνατή εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών γιατί συμφωνώ ότι το πέρασμα από την οδηγία στον κανονισμό ε, από, οδηγία σε κανονισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα έτσι ώστε να εξομαλυνθούν και οι ενδεχόμενες ανομαλίες που παρουσιάζονται λόγω των διαφορετικών κανόνων από χώρα σε χώρα ε, και δεν θέλουμε να παραμείνουν αυτές οι διαφορές γιατί διαφορετικά η κατάσταση θα είναι χαοτική. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και γενικότερα όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να ανασκουμποθούν έτσι ώστε να επιτύχουμε την, μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση. Επίσης, οπωσδήποτε συνοχή με τα άλλα σχετικά ε, θέματα. Ήδη από την αρχή, όταν υποβλήθηκαν οι δύο δέσμες από την Κομισιόν, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλοι οι φάκελοι οι οποίοι βρίσκονται προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπιστούν σε ένα πνεύμα συνολικό έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα ε, μεταξύ των διαφόρων θεμάτων για το κοινό ε, Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου σε εγκάρση, ε, κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Προς ώρας νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας ε, που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας Σε ευχαριστώ. Δεν έχουμε ορίσει κάποια ημερομηνία για την συζήτηση, για την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Μετά τις εκοπές σας ευχαριστώ. Λίγη η πρωινή συνεδρίαση. Τα ξαναλέμε στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ.